Okay. If, we can, uh, if she's not here in 10 minutes... Αν δεν είναι εδώ σε 10 λεπτά, η κυρία Κόνικ θα περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ελπίζω να μπορέσουμε, εντάξει. You don't need to organize that anymore. <laughs> Ήρθε η προσκεκλημένη μας ε, φτάνει από ό,τι φαίνεται, άρα δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Αν είναι σε άλλε συναντήσεις ε, οι συγητές, εντάξει, δεν επήγει. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης ε, που είναι, όπως είχα πει, η παρουσίαση από την Μισελ Κόμνινγκς, πρόεδρο της Eurojust, ε, την οποία καλωσορίζουμε θερμά. Πρόκειται για παρουσίαση της τέταρτης έκθεσης της Eurojust για τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Ο στόχος αυτής της ανταλλαγής απόψεων είναι να μας παρουσιάσει η Eurojust τα ευρήματά της σχετικά με τις εξελίξεις όσον αφορά την ε, αντίδραση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, στο πρόβλημα των αλλοδαπών τροποκρατών μαχητές, μαχητών καθώς και το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στην Μισελ Κόνιγκς και κατόπιν στους ευρωβουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ε, πρόκειται για εφιάλτηση σε το σημερινό πρωινό. Είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμήσει κανείς ε, την κυκλοφορία στις, ε, στο Βέλγιο. Ας ε, προχωρήσουμε λοιπόν στην παρουσίαση της τέταρτης έκθεσης της Eurojust για τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Έχετε λάβει αντίγραφο. Ξεκινήσαμε την ε, εξέταση του θέματος αυτού το 2012 κατά συνάντηση των ε, ειδικών μας ε, για την τρομοκρατία. Το 2012 λοιπόν ε, εντοπίσαμε τα πρώτα σημάδια αλλοδαπών τρομοκρατών μαχητών που επέστρεφαν στο Ιράκ και στη Σύρια για να πολεμήσουν και έκτοτε η σχετική ομάδα έχει επικεντρωθεί κατά 100% σε αυτούς τους μαχητές και την ποινική αντιμετώπιση του θέματος. Το 13, 14, 15 και 16 Ακόμα και ε, στις αρχές αυτού του μήνα ε, έγινε συνάντηση των ε, ειδικών εισαγγελέων για ακριβώς αυτό το θέμα, τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές. Αυτά που σας είπαμε πριν ένα χρόνο ισχύουν ακόμα. Βασιζόμαστε στα ευρήματά μας ήδη από τα πρώτα στάδια των προσπαθειών και ανακαλύπτουμε και νέε πτυχε. Το πρώτο μου λοιπόν μήνυμα είναι ότι η ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία είναι πιο σημαντική από ποτέ, αν θέλουμε να, ε, είμαστε, να έχουμε επιτυχία στον αγώνα μας αυτόν. Και το θέμα αυτό συνδέεται και με τα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο η συγκέντρωση και η ανταλλαγή των αποδεικτικών στοιχείων, ε, είναι Πολύ κρίσιμο είναι και το να συλλέγονται γρήγορα και σε αυτό επικεντρώνονται οι προσπάθειες της Eurojust. Τα στοιχεία είναι θετικά στις επιχειρησιακές μας εργασίες. Έχουμε από την αρχή των προσπαθειών μας έχουμε πολύ καλύτερο συντονισμό τώρα πια και τα μέσα αμοιβαίας αναγνώρισης όπως είναι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και η Ευρωπαϊκή Εντολή Ερευνών που είδε το φως της ημέρας φέτος θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε το στόχο μας. Να <clears throat> συγκεντρώνουμε τα στοιχεία ε, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν εξετάσουμε τα στοιχεία του 2012 και του 2016 όσον αφορά τις έρευνες και τις διώξεις, το 2016 είχαμε 100 33 υποθέσεις σε σχέση με το 2014, όπου είχαμε 33, το 2015 100. Το 2016 λοιπόν 133 υποθέσεις και δικαστικές υποθέσεις που ολοκληρώθηκαν ε, το 2014 180, το 2015 2018 και το 2016 275. Βλέπουμε λοιπόν ε, μια ελαφρά αύξηση στις υποθέσεις ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που δώσαμε στην Europol το 2014, 444 άτομα, το 2015 513 δικάστηκαν και το 2016 580. Το 2016 είδαμε καταδίκες ιδιαίτερα όσον αφορά τους τζιχαντιστές τρομοκράτες. Σε 17 κράτη-μέλη είδαμε ότι το ποσοστό καταδίκηση ήταν εντυπωσιακό. Το 89% των υποθέσεων τελείωσαν σε καταδίκη. Ε, αυτό σημαίνει ότι είχαμε αρκετή επιτυχία όσον αφορά την συλλογή των δεδομένων ε, με σωστό τρόπο σύμφωνα με το κράτος δικαίου. Οι υποθέσεις αυτές ε, οδήγησαν ε, σε φυλάκιση, πρόστιμα, ε, κοινωνική υπηρεσία, εντολές περιοριστικές, καθώς και θεραπεία. Και η μέση ποινή κράτηση στα κρατημέλη ήταν πέντε χρόνια. Όσον αφορά την συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων. Στην περσινή συνάντηση με τους ειδικούς εισαγγελείς επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στα στοιχεία που βασίζονται τις ε, μυστικές πληροφορίες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες πληροφοριών ε, στις ε, διαδικασίες αυτές. Αυτό ήταν ένα ερώτημα που υποβάλαμε στους συναδέλφους και η απάντηση είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες σε κάποιες χώρες. Οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν μπορούν να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία για τις διαδικασίες αυτές. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δηλαδή τα στοιχεία, οι πληροφορίες από τις υπηρεσίες αυτές. Σε άλλα κράτη-μέλη να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για να ανοίξει η διαδικασία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία μόνο εφόσον επιβεβαιωθούν από άλλα ίδια αποδεικτικών στοιχείων. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν θεσπιστεί νόμοι για να ρυθμιστεί η σχέση ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών και τους εισαγγελείς. Καθορίζεται και με ποιον τρόπο θα πρέπει να αποστέλλονται τα αποδεικτικά στοιχεία στους εισαγγελείς. Μπορεί να συμπεριλαμβάνονται σε κάποια έκθεση η οποία θα, θα χρησιμοποιηθεί στη δικαστική υπόθεση και σε άλλες περιπτώσεις ε, μπορούν οι μυστικές πληροφορίες ε, να συμμετάσχουν σε εμπειρογνώμονες ε, στη δικαστική διαδικασία. Συστήνουμε οι δικαστικές αρχές να συμμετέχουν όσο γίνεται νωρίτερα στη διαδικασία, ιδιαίτερα όταν ε, οι πληροφορίες προέρχονται από τρίτες χώρες. Και όταν ενεργούμε στο πλαίσιο της ε, αμοιβαία ε, δικαστικής συνδρομής. Οι πληροφορίε πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με το κράτο δικαίου, θα πρέπει να κρίνονται παραδεκτές στο δικαστήριο και να είναι συγκεκριμένες. σημαντικό θέμα είναι η καταπολέμηση της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Ε, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης αποφάσισαν ότι η Eurojust έχει να παίξει σημαντικό ρόλο στην χαρτογράφηση μέτρων των κρατών μελών ε, για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ πολλές δυνατότητες, ξεκινώντας ήδη με τα πρώτα σημάδια ριζοσπαστικοποίησης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι θέλουν να εγκαταλείψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε σε ζώνες συγκρούσεων, ε, καθώς ε, και την αντιμετώπιση τους όταν ε, επιστρέφουν από αυτές τις ζώνες συγκρούσεων. Σε όλα αυτά τα στάδια υπάρχουν δυνατότητες ε, για παροχή υπηρεσιών στις κοινότητες, ε, να υπάρχουν πολυεπίπεδες διαδικασίες σε επίπεδο εκπαίδευσης, σε σχολείου, οικογένειας, αθλητικών συλλόγων, ε, ακόμα και υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων για να ε, εντοπιστούν και να μετριαστούν τα πρώτα σημάδια της ριζοσπαστικοποίησης. Μόλις δούμε δηλαδή την πρώτη πρόθεση για ε, ριζοσπαστικοποίηση υπάρχει η δυνατότητα να αναλυφθούν βήματα εκτός του τομέα των σοφρονιστικών μέτρων. Κατά την επιστροφή γίνεται ανάλυση κινδύνου, κατηγοριοποίηση των ανθρώπων αυτών και επειδή παρακολουθούμε και την ομολογία και τις ε, δικαστικές υποθέσεις, πριν ε, από την πιθανή καταδίκη εξετάζουμε και το προφίλ κινδύνου για το πρόσωπο αυτό προτού σταλεί στη φυλακή ή αντί για να σταλεί στη φυλακή. Και ακόμα και στη φυλακή υπάρχει πρόβλημα διότι λέγεται ότι ε, είναι οι θερμοκοιτίδες ε, του, της ριζοσπαστικοποίησης οι φυλακές. Αποφεύγεται λοιπόν η συγκέντρωσή τους, χωρίζονται σε διαφορετικές ε, ομάδες. Ε, ή λαμβάνονται άλλα μέτρα για να πετύχουμε την απορριζοσπαστικοποίησή τους, ε, την αποκατάστασή τους. Κάποια κράτη-μέλη ακολουθούν ε, αποκλειστικά την ποινική διαδικασία, εφόσον δηλαδή θεωρηθεί κανείς αλλοδαπός τρομοκράτη μαχητής. Ε, δεν υπάρχει καμία ελεημοσύνη, πηγαίνει κανεί φυλακή σε άλλα κράτη-μέλη, υπάρχουν ε, άλλες προσεγγίσει. Είναι πολύ νωρίς όμω σε αυτή τη στιγμή να έχουμε μελέτη αντικτύπου. Δεν γνωρίζουμε τι θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αλλοδαπών ε, τρομοκρατών μαχητών και την επιστροφή τους με κακές προθέσεις. Ε, ξέρω ότι η Ζουλή Κερχόφεν ε, μαζί με την ε, Eurojust προσπαθεί να εκπονήσει μία πολιτική για τους αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές που επιστρέφουν. Επίσης έχουμε ανακαλύψει ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το αναφέρουμε σε διάφορες εκθέσεις. Βλέπουμε συνεχώς δείγματα αυτής της σχέσης όταν μιλάμε για ε, οργανωμένο έγκλημα, μιλάμε για ε, λαθρεμπόριο όπλων, ε, πλαστογράφηση εγγράφων, εμπορία ανθρώπων ε, ο κατάλογος είναι μακροσκελής. Βλέπουμε όμως ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν αρχίσει να εξετάζουν τη χρήση ειδικών ερευνητικών τεχνικών και εργαλείων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τα χρησιμοποιούν αυτά και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η νομοθεσία βρισκόταν στον πυρήνα της πρώτης έκθεσης Ζητήσαμε ένα αρμονισμένο και πλήρες νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα αυτό έχει γίνει. Έχουμε τη σχετική οδηγία χάρη και στη σκληρή δουλειά του Κοινοβουλίου. Ε, την είδαμε αυτή την οδηγία φέτος τον Μάρτιο που ουσιαστικά Ε, αντιστοιχεί στην απόφαση 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Αυτό είναι πολύ θετικό, διότι είδαμε ότι υπάρχουν κενά στις ποινικέ διώξεις. Είδαμε ότι δεν τιμωρούνται οι επιστρέφοντες αλλοδαπή μαχητές, ε, η εκπαίδευση τους δεν θεωρεί το ε, κολάσιμη πράξη και δεν γίνονταν επαρκείς ε, έρευνες και διώξεις σε διάφορες χώρες. Εξετάζουμε ακόμα την ε, νομολογία και βλέπουμε ακόμα να υπάρχουν κάποιες διαφορές ως προς ε, την ερμηνεία. Σε κάποιες χώρες οι γυναίκες που πηγαίνουν στο Ιράκ και στην ε, Συρία, που μαγειρεύουν, βοηθούν τους μαχητές, τιμωρούνται που στηρίζουν προσπάθειες, δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. Σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό. Το να ε, είναι μια γυναίκα παντρεμένη με έναν μαχητή δεν είναι ε, ποινική πράξη από μόνη της, ε, αλλά υπάρχουν διαφορές και στους επιστρέφοντες δεν βλέπουμε αύξηση του αριθμού, πιθανότερο είναι να μεταφερθούν σε άλλη εμπόλεμη ζώνη, από τη Συρία και το Ιράκ σε άλλο τόπο. Βλέπουμε όμως μια νέα τάση. Βλέπουμε οι γυναίκες και τα παιδιά να επιστρέφουν στην Ευρώπη και χρειάζεται να τους προσέξουμε. Στην πολιτική για τους ε, μαχητές που επιστρέφουν ε, έχουμε συζητήσει ποιος είναι επικίνδυνος, ποιον θα πρέπει να προσέξουμε και με ποιον τρόπο βλέπουμε ότι η τρομοκρατική πρόθεση και η τρομοκρατική δυνατότητα πρέπει να καθορίζει αν κανεί είναι επικίνδυνος ή όχι και δεν θα πρέπει να θεωρείται κανεί μη επικίνδυνος επειδή είναι γυναίκα ή παιδί. Μπορεί να υπάρχει η τρομοκρατική πρόθεση και η δυνατότητα και εφόσον συνεπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία ε, αποτελεί ένα πρόσωπο κίνδυνο. Και ως γυναίκα μπορεί κανείς ε, να έχει ε, τρομοκρατικές δραστηριότητες ε, στο ιστορικό του, οπότε θεωρείται μια γυναίκα επικίνδυνη. Για τα παιδιά είναι πιο πολύπλοκο θέμα. Τα παιδιά που επιστρέφουν ως θύματα θα πρέπει να έχουν πολύ προσεκτική αντιμετώπιση. Επίσης, το ίδιο ισχύει για τους ανηλίκους που επιστρέφουν για να γίνουν μηχανές θανάτου. το ποινικό σύστημα είναι οργανωμένο διαφορετικά σε διάφορες χώρες και αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε στο εγγύς μέλλον. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα θύματα να ε, έχουν φωνή, να ακουστεί η φωνή τους. Και αυτό ήταν το θέμα της φετινής συνάντησης. Ε, πώς θα ασχοληθούμε με τα θύματα μετά από τρομοκρατικές επιθέσεις όπως ήταν ε, οι επιθέσεις ε, στην ε, Γαλλία και στο Βερολίνο. Και φροντίζουμε να μεταδίδουμε τα συμπεράσματά μας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις Σημαντικό είναι να έχουμε συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων με τρόπο γρήγορο. Θα πρέπει όμως να μας αποσχολήσει ε, και ο προϋπολογισμός ε, της Eurojust. Και νομίζω ότι η Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού ασχολήθηκε με το θέμα στην έκθεση για το σχέδιο προϋπολογισμού και έχει ήδη εκφραστεί η ανησυχία. Οι υπηρεσίε τη πρώτη γραμμή, όπω είναι η Frontex και η Europol, έχουν λάβει επαρκή προπολογισμό και επαρκέ προσωπικό. Είμαστε και εμείς σε μέρο ε, αυτών των υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Δεν μπορείτε λοιπόν να σταματήσετε στα μέσα του δρόμου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική και απαραίτητη ε, η συνεργασία και ο συντονισμός σε δικαστικό επίπεδο. Μην σταματήσετε λοιπόν στα μέσα του δρόμου. Εκτιμούμε την στήριξη που μας δώσατε πέρσι, αλλά πρέπει να συνεχιστεί, διότι αυτή τη στιγμή γίνεται όλο και πιο κρίσιμο θέμα. Εάν δεν έχουμε λοιπόν τον απαραίτητο προϋπολογισμό μας για το 2018 και το επαρκές προσωπικό, θα πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερες περικοπές και αυτό θα είναι εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας. Αυτό δεν αποτελεί επιλογή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κόνιξ. Τώρα, οι πολιτικές ομάδες. Η ε, κυρία Ματσόλα βλέπω ότι θέλει το λόγο. αλλά και όποιο άλλο από τι άλλε πολιτικέ ομάδε θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ναι, σα ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την κυρία Κόνιξ που ήρθε και μα ε, παρουσίασε τόσο καλά τι δραστηριότητε τη Eurojust και τις ανάγκες που έχει. Τις ακούμε και να ξέρετε ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά αυτά που ζητάτε. Και χάρηκα πολύ που ασχοληθήκατε και με τα θύματα στην παρουσίασή σας. Για μας είναι ζωτική σημασία. Μερικές φορές, όχι μόνο πιστεύουμε ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασχολούνται αρκετά με τα θύματα όταν συζητούν για τρομοκρατικές επιθέσεις. Γιατί πλήττονται όχι μόνο τα θύματα, αυτά καθεαυτά, αλλά επιπλέον και οι οικογένειές τους, ο περίγυρός τους. Αναφερθήκατε επίσης και στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο διάφορες αρχές αντιμετωπίζουν και μεταχειρίζονται τα δεδομένα που τους φτάνουν, πώς τα επεξεργάζονται. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των αρχών των χωρών μελών. Πώς επεξεργάζονται δηλαδή τις πληροφορίες που τους φτάνουν και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι πληροφορίες και να υπάρχει κάποια συνέχεια, να δίνεται κάποια συνέχεια. Μερικές φορές βλέπουμε ότι η πληροφορία ε, περνάει, αλλά δεν τυχαίνει καμία επεξεργασία. Μετά έχουμε κάποια τρομοκρατική επίθεση και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποια σχέση με τα στοιχεία που είχαμε. Διασυνοριακά Φυσικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να έχουμε τα στοιχεία, αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι η πληροφορία υπήρχε, αλλά δεν κάναμε τίποτα με αυτήν. Άλλος κανείς? Παρακαλώ, κυρία Σύπρο. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα, οπότε δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω όλες τις επεξηγήσεις και τις πληροφορίες που μας έδωσε η προσκεκλημένη μας. Ζητώ συγγνώμη. Όμως, όταν έχουμε να κάνουμε με τους λεγόμενους ολοδαπούς μαχητές, γίνεται πολλή δουλειά. Νομοθεσία, για να δούμε πώς θα εντοπίσουμε τους ε, ριζοσπαστικοποιημένους, πώς θα τους παρακολουθήσουμε, πώς θα παρακολουθήσουμε αυτούς που πηγαίνουν σε τρίτες χώρες, που ενδεχομένως ε, μαθαίνουν πώς να γίνουν μαχητές και μετά επιστρέφουν σε εμά για τρομοκρατικές ενέργειες. Όμως αυτοί οι οποίοι τελικά προβαίνουν σε τρομοκρατικές επιθέσεις, από ό,τι έχουμε διαπιστώσει, είναι ως επιτοπλίστων πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρα κατά τη γνώμη μου δεν φτάνει να παρακολουθούμε τους ανθρώπους αυτούς, να δούμε ποιοι είναι ριζοσπαστικοποιημένοι, να τους παρακολουθούμε και μετά αφού κάνουν την τρομοκρατική ενέργεια να τους βάλουμε στη φυλακή. Μήπως θα ήταν προτιμότερο να δουλέψουμε περισσότερο στην πρόληψη και ακόμα και αν γνωρίζουμε ε, κάποιου ανθρώπου που αρχίζουν να ριζοσπαστικοποιούνται και το μαθαίνουμε αυτό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όχι μόνο να του παρακολουθεί η αστυνομία, αλλά να υπάρξει συνεργασία και με τους κοινωνικά δραστηριοποιούμενους, τις διάφορες κοινωνικές οργανώσεις, ώστε να αποφευθεί συνέχεια. Το έχετε και αυτό υπόψη σας και σε τι βαθμό συνεργάζεστε με άλλες αρχές, κοινωνία των πολιτών κτλ, ώστε να πετύχετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βίνμπερκ και η Ευαζολή βλέπω ότι έχω ζητήσει ακόμα το λόγο. Και η Άννα Γκόμες. Ωραία. Αυτέ οι τρεις και μετά θα επανέλθουμε στην κυρία Κόνιξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να θέσω είναι Πόσα άτομα υπολογίζεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι συνδέονται άμεσα με τρομοκρατικές ε, οργανώσεις. Επίσης αναφερθήκατε σε γυναίκες και παιδιά. Ε, έχουμε νούμερα για πόσους ανθρώπους μιλάμε. Επίσης μιλήσατε για σπαστικοποίηση. Αυτό απαιτεί τεράστιους πόρους. Στη Σουηδία βλέπω τις ανάγκες αστυνομίας. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση στην χώρα μας, ε, διότι έχουμε πολύ λίγους αστυνομικούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους αυτούς που βρίσκονται σε αυτές τις ε, ζώνες κρίσεων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσουμε τη γροθιά μας στο τραπέζι και να δείξουμε σε αυτούς που επιστρέφουν ότι δεν τους επιτρέπουμε την είσοδο στις χώρες μας και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση μαζί τους. Να τους σταματήσουμε. Έτσι νομίζω ότι θα απορριζοσπαστικοποιηθούν πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Εύα Ζουλή. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που ήρθατε για να μοιραστείτε μαζί μας το έργο σας. Βέβαια, δεν μπορώ να πω ότι εικονοποιήθηκα απόλυτα. Θα ήθελα περισσότερες επεξηγήσεις. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το ποσοστό Ευρωπαίων πολιτών στο σύνολο αυτών των ολοδαπών μαχητών. Έχετε κάποια ιδέα ποια είναι αυτή η αναλογία. Και έπειτα, αναρωτιέμαι, όταν χρησιμοποιείται στοιχεία από τις υπηρεσίες πληροφοριών σε μια έρευνα, σε μια διαδικασία, άμα έχουμε να κάνουμε με top secret πληροφορίες, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτές. Αυτές οι πληροφορίες ε, περνάνε και στην άμυνα ή υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ώστε να μπορεί κάποιος να ενημερωθεί και να παρακολουθήσει την κατάσταση. Τέλος, έχετε δημοσιεύσει την τελική έκθεση με ονόματα χωρών μελών. Ευχαριστούμε, Ιάννα Γκόμες. Συγγνώμη, κι εγώ καθυστέρησα λόγω του κυκλοφοριακού, δεν μπόρεσα να σας ακούσω. Όμως το προσωπικό μου ήταν εδώ, οι συνεργάτες μου και θα με ενημερώσουν για το τι είπατε. Λοιπόν, θέλω να αποφελθώ από αυτή την ευκαιρία για να σας ρωτήσω το εξή. Μπορείτε να μας δώσετε τη δικιά σας εντύπωση. Οι χώρες μέλη έχουν προγράμματα για να προωθήσουν την αποφυγή ριζοσπαστικοποίηση ή την άπορη ριζοσπαστικοποίηση, κυρίως στις φυλακές. Εσείς τι συμπεράσματα βγάζετε. Και δεν μιλάω τελικά μόνο για τις φυλακές σε επίπεδο κοινότητας, δεδομένου ότι όλο και περισσότερο γυναίκες ρίζας παστικοποιούνται μέσω διαδικτύου κλπ. Και δεύτερη ερώτηση. Το ότι θα πρέπει να το σταματάμε στα σύνορα είναι γελίο. Είναι το ίδιο όπως ε, κάνουμε όταν λέμε ότι οι μετανάστες και πρόσφυγες ε, είναι τρομοκράτες. Τα προβλήματα με την τρομοκρατία βρίσκονται μέσα στη δικιά μας κοινωνία. Οι περισσότεροι είναι Ευρωπαίοι που έχουν ε, ριζοσπαστικοποιηθεί εξαιτία αποκλεισμού, ηλίθιων πολιτικών, ε, λιτότητας κλπ. Όμως ένα από τα προβλήματα είναι η νομοποίηση του χρήματος που προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες. Είμαστε τώρα στην πέμπτη έκδοση της σχετικής οδηγίας. Οι χώρες μέλη όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αντιστέκονται να εφαρμόσουν την οδηγία για την καταπολέμηση του παράνομου χρήματος που έχει να κάνει και με την καταπολέμηση, την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οπότε εσείς τι συμπεράσματα βγάζετε από τον τρόπο με τον οποίο έχουν αντιδράσει οι χώρες μέλη στην ε, οδηγία αυτή. Και πώς προχωράει. Ακούμε όλο και περισσότερο ότι η τρομοκρατία ε, τελικά με χαμηλό κόστος λειτουργεί και ξέρουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται πολύ συχνά πίσω από, τρομα... από τρομοκρατικές ε, ενέργειες. Οπότε τι συμπεράσματα έχετε βγάλει εσείς που θα μπορούσαμε και εμείς να λάβουμε υπόψη μας τώρα που είμαστε στην ανεθεώρηση της οδηγίας αυτής για την καταπολέμηση του παράνομου χρήματος. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο Μπάτεν και κυρία Φαντφέλτ είδα ότι θέλουν το λόγο, αλλά παρακαλώ ένα λεπτό καθένας, για τελείως δεν θα μπορέσουμε να έχουμε απαντήσεις. Παρακαλώ, κύριε Μπάτεν. Ευχαριστώ χρησιμοποιούμε αυτή την περίεργη διατύπωση μαχητές, λες και είναι ε, παλαιστές ε, βαρέων βαρών. Δεν είναι, είναι τζιχαντιστές. Πρώτα πρέπει να κατανοήσουμε ποιος είναι ο εχθρός μας πριν τον αντιμετωπίσουμε. Και λέτε πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αιτίε, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις βασικές επιπτώσεις. Και το κύριο είναι ότι έχουμε χρήματα που έρχονται από τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και αλλού και ε, χρηματοδοτούν ε, τις ε, ακραίες βαχαμπιστικές σέκτες στα τζαμιά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τουλάχιστον τα μισά τζαμιά χρηματοδοτούνται από έτσι, από εξωτερικού δωρητέ, από τη Σαουδική Αραβία κτλ. Δεν ξέρω αν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία, οικονομικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Ευρώπη. Καλό θα ήταν να έχουμε μια κοινή πολιτική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε και να ε, παρεμποδίσουμε την χρηματοδότηση των ε, τεμενών από εξωτερικέ πηγέ. Ουσιαστικά δηλαδή θα πρέπει όλα αυτά η χρηματοδότηση να έρχεται από το εσωτερικό τη χώρα. Ευχαριστούμε, Νετφέλτ. Ευχαριστώ. Μου κίνησε ενδιαφέρον κάτι που είπε η κυρία Γκόμε για την οδηγία ε, κατά πολέμη νομοποίηση ε, εσόδων με παράνομε πηγέ. Ξέρουμε ότι, για παράδειγμα, η Ουγγρική κυβέρνηση πρόσφατα υιοθέτησε ένα σχέδιο νόμου για τις ΜΚΟ που βασίζεται ακριβώς αυτή την οδηγία για το ξέπλυμα βαρμικού αλλά στόχος είναι ξεκάθαρα να πανοχλήσει ε, και να παρεμποδίσει τη δράση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ξέρουμε και την κατάσταση σχετικά με το κράτο δικαίου στην Ουγγαρία. Αυτό πώ επηρεάζει τη δική σα ε, δουλειά, ποια είναι η εμπιστοσύνη που έχετε στι δικαστικέ αρχέ ε, σε όλα τα κράτη-μέλη και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις ε, ακούστηκαν. Ξέρω ότι είναι αδύνατο ε, να απαντήσετε σε δύο λεπτά. Έχετε λοιπόν λίγο περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας. Αλλά βέβαια πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε και αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Well, I think that uh, those questions were extremely πολύ σημαντικά και επίκαιρα τα ερωτήματα που θίγεται, γιατί ε, εντοπίζεται έτσι και με άλλα σημαντικά στοιχεία. Η καταπολέμηση των λαδοπών μαχητών και του τζιχαντισμού είναι τόσο περίπλοκο ζήτημα που δεν έχει απλές απαντήσεις. Όσο περισσότερες υποθέσεις προσπαθεί κανείς να εντοπίσει και ε, να ασκήσει διώξεις, τόσο πιο πολλά επίπεδα πιθανών λύσεων ε, μπορεί να βρει κανείς. Δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα οι λαδοπιμαχητές, αυτοί δηλαδή που πηγαίνουν στη Συρία και το Ιράκ και επανέρχονται. πραγματικά δεν είναι το μοναδικό θέμα. Οι τελευταίες επιθέσεις είδαμε ότι διενεργήθηκαν από ανθρώπους που δεν είχαν φύγει ποτέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε για μικρούς πυρήνες που κάποιες φορές διασυνδέονται μεταξύ τους, αλλά όχι και απαραίτητα και έχουν κάποιους ε, χαλαρούς δεσμούς με τους αλλοδοπούς μαχητές ε, στις εμπόλεμες ζώνες. Βλέπουμε επίσης ότι η ε, μαζική χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για σκοπούς προσέλκυσης ε, και μελών και χρηματοδότησης για τρομοκρατικούς σκοπούς γίνονται σε αυτά τα βήματα και ότι αυτές οι ενέργειες δεν βλέπουν πάντα το φως της ημέρας γιατί οι χρήστες χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος, το darknet, ε, λειτουργίες κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης. Οπότε έχουμε μία εικόνα κάποιων πλευρών της πραγματικότητας, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι χάνουμε και πολλά. Αν δείτε ότι η χρηματοδότηση γίνεται μέσω ε, διαφόρων μορφών ε, λαθρεμπορίου, έχουμε την αντίληψη ε, ότι ε, χρησιμοποιούνται bitcoins και άλλα εικονικά νομίσματα, οπότε η χνηλάτιση όλων αυτών των πηγών είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε κάποια εικόνα, αλλά όχι την πλήρη εικόνα και το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε τη λύση σε όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό κάπως να χαρτογραφήσουμε ε, τους σκληροπυρηνικούς δηλαδή τέτοιους άλλοδαπες μαχητές. Το ψήφισμα 2322 του ΟΗΕ ε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτόν τον σκληροπυρηνικό μαχητή. Για αυτούς υπάρχει μόνο η καταστολή, δεν υπάρχει άλλη λύση. Για του υπόλοιπου, και έτσι απαντώ σε ένα ερώτημά σα, ίσω υπάρχει καλύτερο τρόπο να αποτρέψουμε ε, τον ακραίο και βίο εξτρεμισμό, να τον καταπολεμήσουμε, να περάσουμε στην απορριζοσπαστικοποίηση και στην επανένταξη στην κοινωνία. Όμως δεν υπάρχει μία λύση για όλους και δεν ξέρουμε όλα τα προβλήματα. Ε, τα τελευταία γεγονότα που είχαμε τρεις επιθέσεις σε τρεις ε, ημέρες, σε τρεις πρωτεύουσες, από άτομα που ποτέ δεν είχαν μπει στο ραντάρ των μυστικών υπηρεσιών, αυτό πραγματικά κάνει τη ζωή μας κόλαση και δεν ε, μας διευκολύνει καθόλου. Για τα στοιχεία που ζητήσατε αριθμητικά δεν τα έχουμε. Αρχίσαμε το 2012 αυτή την προσπάθεια. 7 χώρες το 2012 είχαν δεκάδες τέτοιους ολοδοπούς μαχητές που πηγαίνουν έρχονταν. Και οι, αριθμοί αυξάνονταν συνεχώς. Κάποια στιγμή γινόταν λόγος για 5.000 τέτοια άτομα. Τώρα λέμε ότι δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τεράστιο αριθμό ανθρώπων που θα επανέλθουν και πιστεύω πραγματικά και ειλικρινά ότι τα νούμερα εδώ δεν είναι τα σημαντικά. Το σημαντικό είναι ακόμα να έρθουν και ένας, δύο, τρεις άνθρωποι με ικανότητα και με πρόθεση. Και αυτό μπορεί να ε, φέρει την καταστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ε, Οπότε να μην επικεντρωθούμε σε όλους αυτούς τους αλλοδαπούς μαχητές ε, μόνο, γιατί μπορούμε να έχουμε και ε, ανθρώπους που γεννήθηκαν εδώ και έμειναν εδώ. Ε, μιλούμε και για τους μοναχικούς λύκους, που δεν μου αρέσει βέβαια σαν έκφραση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν αυτούς τους χαρακτηρισμούς του λύκου. Και έχουμε και αυτούς τους πυρήνες. Είναι εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση. Για την κυρία Μέτσολα, για μας θα πρέπει οι αρχέ επιβολή του νόμου, οι μυστικέ υπηρεσίε και οι δικαστικέ αρχέ να ε, δουλεύουν από κοινού. Υπάρχουν ε, ε, πολλέ προσεγγίσει. Γιατί έχουμε ακόμα και πληροφορίες από τις στρατιωτικές αρχές που είναι δύσκολο να περάσουν στο δικαστικό σύστημα. Και αυτό είναι που μελετούμε τώρα, πώς μπορούμε να πάρουμε ε, πληροφορίες από ε, το πεδίο μάχης, να απευθυνθούμε ε, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, σε όσους εργάζονται και χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες στις εμπόλεμες ζώνες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονίες και το καθεξής. Είναι κρίσιμη σημασία σε τα στοιχεία, η συνεργασία με τρίτες χώρες, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Συρία, Λιβύη, Ιράκ. Αυτό βέβαια δεν είναι ο πιο εύκολο τρόπο, όπω καταλαβαίνετε. Πρέπει να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη. Αυτό ακριβώ προσπαθούμε να κάνουμε. Να χτίσουμε ένα δίκτυο σημείων επαφή. Να ε, προσκαλέσουμε την, την αντιπροσωπεία, για παράδειγμα, στην Eurojust για να χτίσουμε την εμπιστοσύνη να βασιστούμε στην ε, διεθνή διασυνοριακή συνεργασία, ε, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης για την ε, συγκέντρωση πληροφοριών. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές στα επιμέρους κράτη-μέλη. Εμείς ως σύσταση λέμε παρακαλούμε να εμπλέκετε και τι δικαστικές αρχές, διασωνερακά δηλαδή τη Eurojust, όσο γίνεται πιο νωρί στη διαδικασία, για να επαληθεύσουμε πώς οι πληροφορίε από τα πεδία μάχης, πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή του, οι μυστικέ υπηρεσίες ή ο στρατός, μπορούν να μεταφερθούν και ε, να διοχετευθούν προ τι δικαστικέ αρχέ με βάση του κανόνε του κράτου δικαίου. I alluded to uh, uh, uh, Μίλησα λοιπόν για τα αποδεκτικά στοιχεία, για το διαδίκτυο μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στη Eurojust πρόσφατα φτιάξαμε και ένα ειδικό εξειδικευμένο ε, δίκτυο και γενικά ε, χρησιμοποιούμε τέτοια δίκτυα. Για το κύβερνο έγκλημα, για παράδειγμα, κάναμε ένα τέτοιο δίκτυο. Δίκτυο για τις γενοκτονίες. Και βλέπουμε ότι σταδιακά ε, συγκεντρώνουμε τέτοιες βέλτιστες πρακτικές, με τα διδάγματα που αντλούμε σε διάφορους τομείς, διασφαλίζουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων αυτών των δικτύων και αυτό κάνει πραγματικά τη διαφορά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μείωση της ριζοσπαστικοποίησης, έχουμε και άλλους τρόπους, όπως ε, το αντιαφήγημα, counter-narrative. Τώρα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, μπορούμε, μάλλον τώρα βλέπουμε ε, ε αφηγήματα που υποκινούν το μίσος και καλούν στη βία. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε το αντίθετο, να δημιουργήσουμε αφηγήματα που ε, διαδίδουν θετικά μηνύματα από ριζοσπαστικοποίησεις και βλέπουμε ότι σε κάποιες χώρες νέοι που επιστρέφουν από εκείνες τις χώρες τραυματισμένοι ε, δεν ε, είναι αυτοί οι σκληροπυρηνικοί επιστρέφοντες και αυτούς μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε σε αυτή την προσπάθεια δημιουργίας ενός αντίθετου αφηγήματος. Και έτσι απαντώ σε όλο αυτό το θέμα ε, της, των άλλων μεθόδων επανένταξη στην κοινωνία μέσω κοινωνική υπηρεσία κ.ο.κ. Μπορούμε να αντλήσουμε έμπνευση από τα όσα βλέπουμε στι ΗΠΑ, στον Ηνωμένο Βασίλειο και στον Καναδά, που υπάρχουν κέντρα από Βλέπουμε ότι και στην πρόληψη του εγκλήματο και στην πρόληψη τη τρομοκρατία έχουμε μια πολυτομεακή προσέγγιση από την ε, περίθαλψη ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, παιδαγωγούς, οικογένειες, οι μάμιδες, όλοι αυτοί προσπαθούν από κοινού να βρουν την ε, καλύτερη και πιο καλά προσαρμοσμένη απάντηση στην ε, απορρισπιστικοποίηση ε, και στην επανένταξη στην κοινωνία. Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα από την κυρία Γκόμες για το ξέπνιμα βρώμικου χρήματος. Ναι, είναι θέμα αυτό. Ήδη το θίξαμε στην πρώτη έκθεση, όπου είχαμε πει ότι αν θέλουμε επιτυχώς να αντιμετωπίσουμε ε, τους ε, τσιχαντιστές τρομοκράτες, πρέπει να ε, παλέψουμε για πλήρης οικονομικές έρευνες. Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να πληρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες και προϋποθέσεις. Υπάρχουν δυσκολίες στην στον εντοπισμό των ε, δραστών για λόγους που έχω ήδη εντοπίσει. Πρόσφατα, σε πρόσφατες ε, καταδίκες κάποιοι καταδικάζονται μόνο και μόνο επειδή έχουν ε, στείλει χρήματα στη Συρία και στο Ιράκ. Δηλαδή, αξιοποιούνται οι ιδιωτικοί τραπεζικοί λογαριασμοί ε, για την χρηματοδότηση ε, τρομοκρατικών ενεργειών των αλλοδοπών μαχητών. Και εκεί και εδώ χρησιμοποιούνται λοιπόν αυτά τα μέσα, αλλά απέχουμε πολύ από το να έχουμε στη θέσή μας όλες τις διασυνδέσεις μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος, εμπορία ανθρώπων, λαθρεμπόριο πολύτιμων μετάλλων και πώς όλα αυτά και συνδέονται με την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Πράγματι, δεν χρειαζόμαστε τεράστιους ε, πόρους, δεν χρειάζεται κανείς τεράστιους πόρους για να ε, διαπράξει μια τρομοκρατική επίθεση, όμως χρειαζόμαστε πόρους για την κατάρτιση, για την διασύνδεση, για, την, για τα ταξίδια που απαιτούνται. Από εκεί δηλαδή είναι σημαντικά αυτά τα οικονομικά στοιχεία. Πρέπει λοιπόν από κοινού να εργαστούμε και να βασιστούμε ε, και στις δικαστικές αρχές και στις αστυνομικές αρχές. Ιδάλλως ε, θα αποτύχουμε. Κυρία Ζωλή, πράγματι αυτή η έκθεση είναι διαβαθμισμένη. Δεν μπορεί να δημοσιευθεί έχει διανεμηθεί σε ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Λάβατε όμως ε, αυτό το, το αντίγραφο της ε, έκθεσης που είναι λοιπόν περιορισμένο και δεν ε, θεωρούμε δεν προβλέπουμε την διάδοση και δημοσίευση μιας τέτοιας διαβαθμισμένης έκθεσης για, για απλούς λόγους αυτή η έκθεση προκύπτει από πολύ συγκεκριμένες και λεπτές ισορροπίες από ε, δικαστές και εισαγγελίες που μας έδωσαν στοιχεία και λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας. Ε, για νομικά και δικαστικά στοιχεία και αν τα μοιραστούμε ή τα δημοσιεύσουμε, αυτό σίγουρα θα έχει αντίκτυπο και στις μελλοντικές δικαστικές έρευνες και υποθέσεις. Οπότε δεν ε, θα άρουμε τον απόρριτο χαρακτήρα αυτής της έκθεσης. Ιδάλλως υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μας. Η εμπιστοσύνη τώρα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι, συνεχώς ε, ε, εργαζόμαστε από κοινού με τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Πρέπει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη με τους ομολόγους μας ε, στις τρίτες χώρες. Δεν ξέρω αν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας, αλλά μπορώ να επανέλθω και να απαντήσω και γραπτός στα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ανταποκριθώ σε αυτήν την πρόσκλησή σα, ε, Θα είναι χρήσιμο για του ευρωβουλευτέ ε, να έχουν πρόσβαση στην έκθεση αυτή, παρότι είναι εμπιστευτική. Υπάρχουν ε, τρόποι επικοινωνίας να το οργανώσουμε αυτό. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο εάν κατόπιν ετήματος των ευρωβουλευτών να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο της έκθεση. Τέθηκαν κάποιες ερωτήσεις ε, σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία. Η κυρία Βίνπερξ ρώτησε σχετικά με το συνολικό αριθμό των ε, μαχητών, ενώ η Εύα Ζολή ρώτησε πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες ε, είναι αλλοδοποί μαχητές. Ίσως θα μπορούσαμε λοιπόν με την με ε, ασφαλή κανάλια επικοινωνία ε, να διαβιβάσετε τα στοιχεία αυτά στη γραμματεία της ΛΥΜΠΕ. Καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορέσετε να απαντήσετε αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις εδώ στην δημόσια συζήτηση. Νομίζω όμως ότι θα είναι χρήσιμο και για τις μεταξύ μας σχέσεις ε, να μπορέσουν να μεταφερθούν οι πληροφορίες κατευθείαν στους ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ζητώ συγγνώμη Λυπάμαι μάλλον που δυσκολευτήκατε να καταστάσετε. Ελπίζω να μπορέσετε να αποχωρήσετε πιο ανώδυνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς δεν ήμουν η μόνη που είχε κολλήσει στην κίνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλημέρα. Okay, dear colleagues, we will have to... Συνάδελφοι, πρέπει να προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, που είναι η παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ε, προτινόμενης οδηγίας ε, για την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου. Παρουσιάστηκε το Δεκέμβριο του 2016 και βασίζεται στην ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε και τις ε, συστάσεις ε, της ειδική ομάδας ε, χρηματοοικονομικής δράσης. Δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη μέλη αυτής της ομάδας. Η πρόταση αυτή πηγαίνει ακόμα πιο πέρα όσον αφορά τον αριθμό των αδικημάτων σχετικά με την καταπολέμηση της νομοποίησης εσόδων, όσον αφορά την αποσύνδεση ε, της ε, νομοποίησης παράνομων εσόδων από την ε, καταδίκη για εγκληματική δραστηριότητα. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την πρώτη του γενική προσέγγιση στις 8 Ιουνίου του 2017. Θα δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρουσιάσει σύντομα την πρόταση αυτή και κατόπιν στον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και κατόπιν σε άλλους ευρωβουλευτές. Δίνω λοιπόν καταρχά ε, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει το σχέδιο οδηγίας της. Παρακαλώ. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο παρακαλώ ή χρησιμοποιήστε κάποιο άλλο μικρόφωνο. Μήπως απλά να αλλάξετε θέση. Συγγνώμη αλλά νομίζω ότι έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Ελπίζω να λειτουργεί τώρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ κύριε Άλπρεχτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτήν την πρώτη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. που αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινοτική ε, αντίδρασης ε, στην νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας. Ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης ε, για την καταπολέμηση τη τρομοκρατίας που υιοθετήθηκε πέρσι. Συμπληρώνει το προληπτικό πλαίσιο το οποίο αναθεωρείται αυτή τη στιγμή. Το πλαίσιο αυτό καθορίζει τους κανόνες σχετικά με την υποβολή αναφορών ε, για ύποπτες ε, συναλλαγές και στόχο έχει να αυξήσει την διαφάνεια στις ε, οικονομικές συναλλαγές. Και η πρόταση που σας παρουσιάζουμε σήμερα έχει να κάνει με την αντίδραση από πλευράς ποινικού δικαίου. Στόχος λοιπόν είναι να ενισχύσουμε το ισχύον πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομοποίησης εισόδων εισάγοντας ελάχιστους κανόνες, ορίζοντας το αδίκημα της νομοποίησης εσόδων ε, και καθορίζοντας ε, και τις ποινές. Στόχος είναι φυσικά να βελτιώσουμε τη διασυνοριακή συνεργασία και να αποτρέψουμε ε, τρομοκρατικές δραστηριότητες και ο τελικός στόχος είναι να βελτιώσουμε την εσωτερική ασφάλεια και την ασφάλεια των πολιτών μας. Η νομοποίηση παράνομων εσόδων επιτρέπει σε εγκληματικέ οργανώσεις να επωφεληθούν από τις ε, παράνομες δραστηριότητές τους και να συνεχίσουν τις λειτουργίες τους. Έτσι αποτελεί σημαντική συμβολή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος η συγκεκριμένη πρόταση. Όπως άλλωστε ακούσαμε και από την πρόεδρο τη Eurojust. Το Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν στα 2,1 τρισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα από εγκληματικέ δραστηριότητε, ε, συνολικά δηλαδή το 3,6% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσό των χρημάτων ε, που παράγονται από παράνομες δραστηριότητες υπολογίζεται σε 110 δισεκατομμύρια το χρόνο, κάτι που αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να επωφεληθούν πλήρως ε, οι εγκληματίες από ε, τα προϊόντα των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων θα πρέπει να μοποιήσουν τα έσοδα. Το παρόν ε, πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι ούτε πλήρως ε, ούτε συνεκτικό για να μπορεί να είναι και απόλυτα αποτελεσματικό. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν ποινικοποίησει την νομιμοποίηση εσόδων. Υπάρχουν όμως ακόμα σημαντικές νομικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Οι διαφορές αυτές δημιουργούν εμπόδια που όπως υπόθηκε, εμποδίζουν την διασυνοριακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η νομιμοποίηση των εσόδων. Οι διαφορές αυτές, ε, τις διαφορές αυτές εκμεταλλεύονται οι εγκληματικές οργανώσεις. Η οδηγία λοιπόν στόχο έχει να εξαλείψει τα εμπόδια αυτά, ε, δημιουργώντας κοινό ορισμό της νομιμοποίηση εσόδων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζει, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, μία διεθνή υποχρέωση ε, που απορρέει από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την ε, ομάδα δράσης του ΩΣΑ. Η οδηγία πηγαίνει πέρα από αυτές τις απαιτήσει, καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο κυρώσεων και ποινικοποιεί και την νομοποίηση εσόδων από το ίδιο πρόσωπο. Δηλαδή, ε, η νομοποίηση γίνεται από το ίδιο πρόσωπο που έκανε και την εγκληματική ενέργεια. Βλέπουμε ότι οι εγκληματίες γενικά νομοποιούν μόνοι τους ε, τα έσοδα από τις ε, δραστηριότητές τους και θέλουμε να ποινικοποιήσουμε αυτό ακριβώς. Ε, ε, ε, στην προηγούμενη στην προηγούμενη παρουσίαση ακούσαμε για τις εγκληματικές δραστηριότητες που παράγουν χρήμα το οποίο κατόπιν νομιμοποιείται και σε διεθνές επίπεδο απαιτείται από τις χώρες να καλύπτουν τουλάχιστον 21 κατηγορίες εγκλημάτων από την εμπορία ανθρώπων μέχρι την απάτη, το οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θεσπίζει έναν τέτοιο ελάχιστο κατάλογο, προσθέτει όμως εδώ το κυβερνοέγκλημα. Το κυβερνοέγκλημα αποτελεί απειλή στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, απειλή στην οικονομία, απειλή για την επιτυχία της ε, ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος του κυβερνοεγκλήματος στα δικαιώματα των πολιτών και τα διάφορα οικονομικά συμφέροντα. Πρόεδρε, Κλείνοντας, ε, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να κλείσουμε τα κενά αυτά που έχουμε εντοπίσει. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο εκτιμάει ότι είναι απαραίτητο να ενεργήσει γρήγορα και να καταλήξουμε σε ε, λύση εντός του μήνα. Επικροτούμε το ξεκίνημα της συζήτησης στο Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι και εσείς θα μπορέσετε να καταλήξετε σύντομα σε μια λύση που θα επιτρέψει να ξεκινήσουν οι διαθεσμικές ε, συζητήσεις. Και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μέχρι το τέλος της χρονιάς. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Κοράου, ο εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ακριβώς όπως υπενθύμησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κλιματική δραστηριότητα υπάρχει, υφίσταται, για να οδηγήσει σε κέρδη, σε ωφέλη, σε κέρδη, από τα οποία μπορεί να αποφεληθεί κανείς μόνο εφόσον υπάρξει νομιμοποίηση των ε, εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Έχουμε να κάνουμε εδώ με ένα κατακαιρματισμένο βέβαια τοπίο όσον αφορά τις διάφορες διατάξεις. Καλό είναι λοιπόν που μπορούμε να δράσουμε. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές όσο γίνεται καλύτερα. Από τη δικιά μου την πλευρά έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τη διαδικασία αφενός αλλά και όσον αφορά την ουσία αφετέρου. Επί της διαδικασίας. Η πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σίγουρα είναι καλή. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση εκκίνησης. Βέβαια υπήρξε ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή, μόνο την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε στα χέρια μας μια εσωτερική μελέτη που είναι απόρριτη, μελέτη ε, την οποία δεν μπορούμε να τη δώσουμε στους δικούς μας εμπειρογνώμονες σε εθνικό επίπεδο. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να είχε γίνει μια μελέτη αντικτύπου. Δεν ξέρω. Εν πάση τώρα μας πιέζουν, μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε γρήγορα. Εγώ δεν συμφωνώ. Συνεπώ, εμείς θα αρκεστούμε σε αυτήν την μελέτη και θα προσπαθήσουμε ε, να τα καταφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα. Έρχομαι τώρα στην ουσία. Υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε. Θα ακούσουμε εμπειρογνώμονες και αυτό θα το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Για το θέμα αυτό ακριβώς της νομιμοποίησης εσόδων. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το τι συμβαίνει. Και μετά υπάρχει και το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Και εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο και έπειτα υπάρχει και το θέμα της κατηγορίας των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στην οδηγία αυτή. Όταν μιλάμε για ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις, πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει αναρμόνιση των κυρώσεων. Και εδώ πρέπει να μπούμε περισσότερο στο βάθος για να βρούμε τη σωστή απάντηση. Πάντως, όπως το έχω ήδη πει, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς. Έχω ήδη συναντηθεί με τους κοιόδες εισηγητές και όπως σας είπα θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε όσο γίνεται καλύτερα στο κοινοβουλευτικό αυτό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Τι σκιώδη συζητητές θέλουν τώρα το λόγο, οι άλλοι ευρωβουλευτές, παρακαλώ. Η Μόνικα Χολμάγερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Πιστεύω από την πλευρά μου ότι αυτό το πλαίσιο το οποίο μας παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που με συναπόφαση αποφασίζεται και που δεν έχει αποφασίσει ακόμα το Συμβούλιο, θυμίζει άλλες κατευθυντήριες γραμμές και το περιεχόμενο μοιάζει πολύ. Πάντως υπάρχουν κάποια πράγματα εδώ που δεν είναι απλά αυτό το θέμα ε, της νομιμοποίησης που γίνεται από τον ίδιο τον εγκληματία Νομίζω ότι είναι καλό να ακούσουμε και πραγματογνωμοσύνη από τη Eurojust και νομίζω ότι αυτό το έχουμε προβλέψει. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα ε, και άλλα, στο οποίο αναφέρθηκε και η κυρία Γκόμες χτες. Γιατί μερικές φορές δεν υπάρχει τιμωρία γιατί το αδίκημα στη χώρα όπου αυτό έλαβε χώρα δεν οικοποιείται. Και άρα με ένα τιμόρυτο. Η έλλειψη δικαστικής συνεργασίας λοιπόν μεταξύ των χωρών μελών είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει πάρα πολύ στον χώρο, στα δικήματα που γίνονται στον χώρο. Και αυτό πρέπει να το καλύψουμε. Λοιπόν, στη Γερμανία 12 δισεκατομμύρια ε, ήταν η απώλεια από την τελευταία επίθεση που είχαμε στον κυβερνοχώρο. Εδώ μιλάμε λοιπόν για 12 δισεκατομμύρια. Το φαντάζεστε. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να δούμε τελικά τι γίνεται και με τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά τα οποία βγήκαν από την Κεντρική Τράπεζα και χρησιμοποιήθηκαν ε, μέσω διαφόρων ε, διόδων σε παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την εναρμόνιση, πράγμα που σημαίνει ότι αν στις διάφορες χώρες μέλη ε, κάποια επαγγελματική πράξη δεν τιμωρείται, γιατί αυτά ψάχνουν και οι εγκληματίε να βρούνε πού υπάρχουν κενά στην νομοθεσία και υποφελούνται από αυτό και τα καταφέρουν και πάρα πολύ καλά. Κυρίω όταν μιλάμε για τέτοια χρήματα, δισεκατομμύρια. Γι' αυτό και λέω ότι πρέπει να υπάρξει αναρμόνιση ώστε να μην υπάρχουν πια τέτοια κενά. Και εμείς θα φροντίσουμε να προχωρήσουμε. Το χρονοδιάγραμμα του εισηγητή είναι πολύ καλό πιστεύω. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ιάννα Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για πολύ σημαντική δουλειά. Η εναρμόνιση δηλαδή των κυρώσεων από πλευρά των χωρών μελών κάθε φορά που έχουμε νομοποίηση εσόδων από εγκληματικέ δραστηριότητε. Και δεν πρόκειται εδώ πέρα μόνο για την ε, αναθεώρηση της πέμπτης οδηγίας, αλλά πρόκειται και από τι έρευνε που κάνουμε όσον αφορά τα Panama Papers, τα έγγραφα του Παναμά, έτσι στην ε, αντίστοιχη επιτροπή. Πολλά πράγματα πρέπει να εναρμονιστούν στην Ευρώπη. Η ποινικοποίηση των εγκλημάτων αυτών, για παράδειγμα, είναι κάτι απολύτως αναγκαίο αν θέλουμε να είμαστε και αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος και των συναφών οργανωμένων εγκλημάτων. Βέβαια το βασικό είναι η πολιτική βούληση. Χτε, όπω και άλλοι συνάδελφοι, έφυγα κατά τις 9 μετά από 6 ώρε που δουλεύαμε πάνω στην πέμπτη οδηγία, η οποία τελικά μάλλον θα περάσει στην επόμενη Προεδρία, γιατί οι χώρες μέλη αντιστέκονταν. Για τρει ώρες ήμασταν εκεί και περιμέναμε. Τι θα κάνουν οι χώρες μέλη οι οποίες έπρεπε να αποφασίσουν για πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορούσε να δεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα τρας. Φυσικά, δεν μπορείς να παριστάνεις ότι καταπολεμάς αυτό το έγκλημα όταν υπάρχουν τεράστια κενά στις νομοθεσίες των χωρών μελών για τα τρας, για διάφορα ιδρύματα κλπ δεν υπάρχει έλεγχος επειδή λένε α, αναλογικότητα, προστασία, ιδιωτικότητα και δεν συμμαζεύεται. Αλλά, εν πάση παρά τις πολιτικές αντιστάσεις ορισμένων χωρών μελών, υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Αυτό το σύστημα καταπολέμησης της νομοποίησης παράνομου χρήματος έχει να κάνει με την έννοια που λέει ότι πρέπει να καταγγέλλεται κάθε ύποπτη κίνηση που εμπίπτει στην προσοχή τραπεζών ή ξέρω εγώ ποιον άλλον. Αλλά το πρόβλημα είναι, και εμείς το βλέπουμε αυτό και στην Επιτροπή για τα Έγγραφα του Παναμά, ότι οι περισσότερες από αυτές ε, τις οντότητες που είναι υποχρωμένες να καταγγείλουν τέτοια φαινόμενα δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν απλά. Οι περισσότεροι από αυτούς που το κάνουν τελικά είναι η τράπεζα για τα χρήματα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι σύμβουλοι δεν το κάνουν. Δεν καταγγέλνουν, δεν νιώθουν ότι οφείλουν να το κάνουν. Οπότε αυτό είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας. Και ούτε το κάνουν και οι εποπτικές αρχές, δεν καταγγέλουν οι κεντρικές τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές κλπ. Αυτή είναι η πρώτη δυσκολία. Και η σύνδεση βέβαια με τους παραλογικούς παραδείσους είναι προφανής. Πάνε τα χρήματα εκεί στους φορολογικούς παραδείσους και μετά όταν επιστρέφουν επενδύονται σε σπίτια κλπ. Και, και κανένα πρόβλημα. Έπειτα υπάρχει το predicate offense. Το κύριο αδίκημα. Ποιε είναι οι επιπτώσει Στη χώρα μου, την Πορτογαλία, πρόσφατα είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση από ένα εφετείο κατά απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που είχε πει ότι μια τέτοια έρευνα για νομιμοποίηση παράνομου χρήματος δεν μπορεί να γίνει. Είχε να κάνει με τον αντιπρόεδρο της Αγγόλα γιατί το κύριο αδίκημα, διαφθορά ή ξέρω εγώ οποιοδήποτε άλλο, δεν έλαβε χώρα στην Πορτογαλία αλλά στην Αγγόλα. Οπότε παρά τι αποδείξει που υπήρχαν ότι το παράνομο χρήμα είχε μπει στην Πορτογαλία, το κύριο αδίκημα δεν μπορούσε να διερευνηθεί στην Πορτογαλία. Τελικά το εφετείο έτρεψε την απόφαση αυτή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου και είπε ότι παρά το γεγονό το κύριο δίκημα έλαβε χώρα στην Αγγόλα, η Πορτογαλία μπορεί και θα έπρεπε να ερευνήσει το αδίκημα τη νομοποίησης παράνομου χρήματος. Αναφερθήκαμε και στα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Τα περισσότερα από αυτά λαμβάνουν χώρο χωρίς καν να αντιλαμβανόμαστε ότι λαμβάνουν χώρο τα bitcoin, το εικονικό χρήμα, το fintech που ονομάζεται τώρα που είναι χρηματοπιστωτική τεχνολογία. Χρειαζόμαστε εμπειρογνώμονε για να διαρευνήσουμε τέτοια ζητήματα. Τέλος, για τις κυρώσεις. Αυτό που μαθαίνουμε από τα έγγραφα του Παναμά είναι ότι ό,τι κυρώσει και αν βάλει στην νομοποίηση του παράνομου αυτού χρήματο από κλιματικέ οργανώσεις, φυλακές, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι τίποτα. Εδώ είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε. Και θα ολοκληρώσω με το ότι πρέπει να έχουμε ακράσει με τη Eurojust, τη Europol, με το FIUs, προκειμένου να μάθουμε τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν και αυτοί, προκειμένου αυτή η τόσο ουσιαστική οδηγία να μην χάσει ακριβώς την ουσία της. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Να είσαστε λίγο πιο σύντομοι την επόμενη φορά, αλλιώ πραγματικά θα έχουμε πρόβλημα με το χρόνο σήμερα. Ωραία. Επόμενος σκιώδη. Ε, ο κύριο Γέζεκ είπε ότι θέλει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω αυτή την πρόταση που, όπως έχει διπωθεί, εξηγεί και γιατί απέτυχε ο χθεσινός τριμερής διάλογος για την πέμπτη οδηγία για την νομοποίηση όταν με παράνομε πηγές. Ε, πάντα ε, εμεί ζητούμε περισσότερη διαφάνεια, το Συμβούλιο όμω μας ε, παρεμποδίζει. Ανέφερε η Άννα και τις εργασίες της Επιτροπής για τα έγγραφα του Παναμά, ειδικά στη φορά τη διασυνοριακή διάσταση της ε, καταπολέμησης νομοποίησης εσόδων με παράνομε πηγές. Καλό είναι συμπληρωματικά να εντοπίσουμε και να εξαλείψουμε ε, διαφορές ε, στο νομικό καθεστώς ε, των πρώτων μελών και να υπάρξει μια εναρμόνιση ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το Συμβούλιο έχει ήδη ε, υιοθετήσει αυτή τη γενική προσέγγιση και είπε και ο εισηγητής ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ε, μια καλή αφετηρία και εγώ συμφωνώ με αυτή τη γνώμη καθώς δεν είναι και τόσο μακροσκελής η πρόταση, νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε αρκετά γρήγορα, χωρίς να υποτιμούμε τον χρόνο που απαιτείται ή τη σημασία του θέματος. Νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε γρήγορα και ε, να λειτουργήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά για να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση των συντομότερων δυνατών. Ευχαριστώ. Η Εύα Ζολή. Και μετά η κυρία Τσινίτση και πρέπει να κλείσουμε μετά τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση πραγματικά είναι απίστευτη γιατί το σύνολο των κρατών μελών ε, συμμετέχουν και στη ΚΑΦΗ και εδώ και 30 χρόνια η διεθνής κοινότητα ε, προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτό το φαινόμενο. Ξέρουμε λοιπόν τις αδυναμίες και πραγματικά έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τη δική της δεσμευτική οδηγία. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό, αυτή η μαύρη τρύπα μέχρι τώρα, είναι ότι σε πολλές χώρες η φοροδιαφυγή δεν ε, θεωρεί το τέτοιο κύριο αδίκημα. Και έτσι είχαμε ένα τεράστιο χάσμα. Ε, η οδηγία λοιπόν θα πρέπει να διευκρινίζει ότι το σύνολο των αξιόπινων πράξεων ε, που ε, τιμωρείται με ένα έτος φυλάκισης και παραπάνω μπορούν να θεωρηθούν να επιτείνουν ε, ε, περαιτέρω, να περαιτέρω ποινή σε σχέση με τα αρχικά δικήματα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τσινίτσι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους σκιώδης εισηγητές που έκαναν πάνω σε αυτήν την πολύ σημαντική οδηγία. Πρόκειται για οδηγία που περιμένουμε με ανυπομονησία, διότι έχουμε μεν άλλες οδηγίες, χρειαζόμαστε όμως μία που να εξετάζει τα μέσα του ποινικού δικαίου για την αντιμετώπιση αυτού του είδους των εγκλημάτων. Πρόκειται λοιπόν για οδηγία μεγάλης σημασίας. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι εργασίες όσο γίνεται πιο γρήγορα χωρίς όμως ε, αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε διαστικά. Η νομιμοποίηση των εσόδων ε, από το ίδιο το πρόσωπο που έχει διαπράξει το πρώτο έγκλημα είναι ένα θέμα που στην Ιταλία έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα στην καταπολέμηση Τη εγκληματικότητα, διότι συχνά πίσω από την ομοποίηση των εσόδων κρύβονται ε, σημαντικά ε, σοβαρά εγκλήματα. Τώρα λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε ευρωπαϊκή προσέγγιση στο θέμα αυτό και όπως ήδη ακούσαμε, η συνεργασία, ο συντονισμός κατά τις έρευνες από πλευράς ε, των αρχών είναι πολύ σημαντική. Πάντα βρισκόμαστε ένα βήμα πίσω από τους εγκληματίες. Πρέπει όμως όσον αφορά για παράδειγμα το κυβερνοέγκλημα θα πρέπει να επιταχύνουμε διότι γνωρίζουμε ότι το οικονομικό έγκλημα σήμερα περνάει μέσα από το διαδίκτυο. Δύο πτυχές θα ήθελα να επισημάνω. κατά τη γνώμη μου, ακόμη δεν έχουμε κοινό ορισμό των εγκληματικών οργανώσεων, διότι όπως είπα πριν, ε, συχνά τέτοιου είδους ε, εγκλήματα κρύβουν από πίσω τους σε μια εγκληματική οργάνωση. Έχουμε μεν έναν ορισμό, δεν είναι όμως αρκετά σαφής, διότι δεν έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο όλα τα κράτη-μέλη αυτές τις διατάξεις ή τις έχουν μεταφέρει με διαφορετικό τρόπο. Τώρα λοιπόν χρειαζόμαστε κοινή έννοια, κοινό ορισμό για τις εγκληματικές οργανώσεις και να πρόκειται για δεσμευτικό ορισμό. Αυτό θα αποτελέσει η βάση και για όλες τις άλλες οδηγίες που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο. Μου ζητήσατε να είμαι σύντομη, γι' αυτό θα κλείσω λέγοντας ότι το άρθρο 10 στο έγγραφο της ανακοίνωσης δεν περιέχει ελάχιστο κατάλογο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε κάτι τέτοιο, διότι έχουμε εγκληματικές οργανώσεις και θα είναι πολύ χρήσιμο να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στη συγκεκριμένη οδηγία. Διότι Γίνονται διαφόρων ειδών έρευνες όπως είναι ε, οι υποκλοπές ε, τηλεφώνων κλπ. Ε, θα πρέπει όμως να εργαστούμε περισσότερο πάνω στο θέμα του συντονισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν πάνω στο θέμα αυτό, διότι το χρειαζόμαστε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος θα πάρει το λόγο ο εισηγητής ε, και ίσως μπορεί να μας δώσει και μερικές πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου έκθεσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χτες αποφασίσαμε Αποφασίσαμε λοιπόν να επιταχύνουμε κάπως την ε, κίνηση δηλαδή να επιταχύνουμε λίγο το χρονοδιάγραμμα και να έχουμε την έκθεση αυτή τέλη Σεπτεμβρίου. Το Σεπτέμβριο θα έχουμε λοιπόν συναντήσεις με εμπειρογνώμονες για τις τροπολογίες μέσα Οκτωβρίου θα είναι η προθεσμία. Άρα τέλη Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και έτσι θα μπορέσει να κλείσει αυτή η υπόθεση το Νοέμβριο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε και θα περάσουμε αμέσω στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη που είναι παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το 2016 του Στέφαν Κέσλερ που είναι πρόεδρος του Συμβουλευτικού Φόρουμ του Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, πολιτικές και ανώτερος πολιτικός και νομικός σύμβουλος επίσης στην υπηρεσία εισιτών για τους πρόσφυγες και τον Ντέις Κοτζούλε, αξιωματικός ε, σύνδεσμος επίσης της ε, Υπηρεσίας για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Αθηνών για τη Frontex, εξ ονόματος της Σουφιάν Ατζάλη, πρόεδρος του Βουλευτικού Φόρουμ της Frontex για θεμελιώδεις δικαιώματα. Για ελάτε εσείς εδώ. Για το επόμενο θέμα, όπως σας είπα, έχουμε προσκαλέσει δύο οργανώσεις που συμμετέχουν στο Συμβουλευτικό Φόρουμ για την Frontex για να μας παρουσιάσουν τις δραστηριότητες του σώματος. Ε, έκθεση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα. Ο Στέφαν Κέσλερ είναι δίπλα μου για τους πρόσφυγες και ο κύριος Κοζούλε από την ύπατη αρμοστεί για τους πρόσφυγες. Δέκα λεπτά, όπως θέλετε το μοιράζετε. Και μετά θα ακούσουμε ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές μας. Θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, ερωτήσεις για να απαντήσετε. Τώρα όμως, σας παρακαλώ, την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να συζητήσουμε μαζί σας την τέταρτη αυτή έκθεση του Συμβουλευτικού Φόρουμ της Frontex για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα σύνορα. Δέκα λεπτά μας δώσατε για την παρουσίαση αυτή και θα προσπαθήσω, γιατί ξέρω ότι είναι Γερμανός ο Πρόεδρος, να τηρήσω το χρόνο μου. Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε έξι σημεία της έκθεσης αυτής και να καταλήξω σε κάποιες παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν ναι, με τη συζήτηση που γίνεται όσον αφορά τη διάσωση στη θάλασσα. Πρώτον λοιπόν, το φόρουμ μας συμμετείχε στις συζητήσεις για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ρύθμισης του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή. Δυστυχώς, Περισσότερες από τις συστάσεις μας δεν έχουν συμπεριληφθεί στην νομοθεσία αυτή. Έτσι, λοιπόν, κάναμε διάφορες συστάσεις στη Frontex, προκειμένου να υπάρξει ένας μηχανισμός στη Frontex για ατομικές προσφυγές. Και έτσι όπως ε, έχει σήμερα το πράγμα, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι επαρκής, δεν είναι ικανοποιητικός για να διασφαλίσει πρόσβαση σε διόρθωση εφόσον υπάρχουν προσφυγές για κακή δίκηση. Το φόρουμ μας επίσης είπε ότι οι κανόνες που διέπουν το μηχανισμό αυτό θα έπρεπε να μην αρκούνται στο άρθρο 72 του κανονισμού, αλλά να πηγαίνουν πιο μακριά. Μεταξύ άλλων, θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς τηρούνται οι κανόνες επί της διαδικασίας, να διευκρινίζεται το χρονοδιάγραμμα επίσης της διαδικασίας επεξεργασίας των προσφυγών και να υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγών να γίνονται ανώνυμα. Όμως δεν έγινε αυτό. Και επαναλαμβάνουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει και περισσότερο προσωπικό που να είναι στην υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το έχουμε πει αυτό από την αρχή, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε. Χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Οι συστάσεις μας, οι μας πιστεύουμε ότι εξακολουθούν να ισχύουν. Και ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξη της δικιάς σας Επιτροπής απέναντι στη Frontex για αυτά. για να υλοποιηθούν οι συστάσεις μας αυτές. Το δεύτερο είναι ότι χαιρόμαστε που υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πουλ που θα ελέγχει τις επιστροφές. Θα παρακολουθεί δηλαδή τις διαδικασίες επιστροφής των ανθρώπων. Επιμένουμε ότι αυτή η ελεγχή πρέπει να γίνονται ανεξάρτητα. Το πουλ αυτό να είναι ανεξάρτητο δηλαδή για όλες τις περιπτώσεις επιστροφών, αναγκαστικών επιστροφών. Αλλά μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος στις επιστροφές αυτές, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες επιστροφών έλεγχος από ανεξάρτητους. Τρίτον, συζητάμε με την Frontex για τη συνεργασία της με τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένα λεπτό ζήτημα. Η Τουρκία αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο μεγάλη σημασία έχει μια τέτοια συνεργασία. Ε, κατάρτιση επίσης της Λιβικής ακτοφυλακής είναι ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει πόσο λεπτό και δύσκολο είναι το ζήτημα της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Τέσσερα. Το φόρουμ μας έχει δουλέψει για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Frontex. Στηρίζουμε το θέμα αυτό της προστασίας των παιδιών από πλευράς της Frontex και πρέπει να επεκταθεί. Έχουμε αρχίσει συζήτηση για μελέτη όσον αφορά την υποχρέωση διάσωσης των παιδιών. Τα αποτελέσματα μας έχουν βοηθήσει να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που υποβάλλουμε στην Frontex και ελπίζουμε ότι έχει αρχίσει μια καρποφόρα συζήτηση με τη Frontex για την διαχείριση των συνόρων όσον αφορά την προστασία των παιδιών. 5. Συνεισφέρουμε στην αναθεώρηση της στρατηγικής της Frontex για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενσωματώνοντας τα πορίσματα της αξιολόγησής μας όσον αφορά την ε, διάσταση του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες της Frontex. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε για την αναθεώρηση της στρατηγικής ε, αυτής της Frontex μέσα στο 2017 και ο τελικός στόχος θα πρέπει να είναι μια στρατηγική θεμελιδών δικαιωμάτων που να αντικατοπτρίζει την εντολή της Frontex και να την ενισχύει Υπήρξε εντολή για την ενίσχυση της εντολή της, τώρα η στρατηγική που θα ακολουθήσει θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην αυτή εντολή για την ενίσχυση των τίτων της. Και το έκτο που θέλω να αναφέρω είναι ότι το φόρουμ μας έχει συνεισφέρει στην εκπόνηση και στην ε, εφαρμογή κατάρτισης με συγκεκριμένο υλικό. Εδώ πρέπει να υπογραμμίσω τη σημαντική δουλειά που έχει γίνει και που υιοθετήθηκε τον Ιούνιο που μας πέρασε. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με μία προσωπική παρατήρηση για την συζήτηση που γίνεται σήμερα όσον αφορά τη διάσωση. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ...2005 πρόσφυγες και μετανάστες έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο. από την 3η Ιανουαρίου φέτος του 2017 μέχρι τις 23 Ιουνίου. Διάφορε μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν ε, οργανώσει δραστηριότητε διάσωσης προκειμένου να αποφύγουν περισσότερους ακόμα θανάτους. Όμως, κάποιοι αξιωματούχοι της Frontex έχουν ε, πει πράγματα στα μέσα ενημέρωσης που μπορεί κανείς να τα εκλάβει σαν κατηγορία από πλευρά της Frontex απέναντι στις ε, μη κυβερνητικέ αυτές οργανώσεις που έχουν διασώσει κόσμο. Θέλουμε λοιπόν η Frontex να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Και χαιρόμαστε που η Frontex το έκανε πολύ πρόσφατα με επιστολή προς τους ευρωβουλευτές εδώ, λέγοντας ότι οι μη κυβερνητικές αυτές οργανώσεις κάνουν αυτό που ακριβώς πρέπει να κάνουν, να σώζουν τις ζωές των ανθρώπων. Αν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις δεν δραστηριοποιούνταν, τότε ακόμα περισσότεροι πρόσφυγες και μετανάστες θα είχαν χάσει τη ζωή τους. Συνεπώς, υπενθυμίζουμε στην Επιτροπή σας ότι πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να οργανωθούν ασφαλείς δίωδοι εισόδου των προσφύγων και μεταναστών για να μην πρέπει να χάνονται έτσι ζωές στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you Ευχαριστώ. Εσείς κάνατε την παρουσίαση και η συνάδελφός σας θα απαντήσει στους ευρωβουλευτές. Ναι, και οι δύο. Λοιπόν, τέσσερα μέλη, πέντε έχουν ζητήσει το λόγο. Κυρία Γκόμες, Σπινέλη, Άντρισον, Ρίσπρεκ και Βεργιά. Η κυρία Εντφέλτ. Κύριος Κρίστα. κυρία Τσινίτση. Εντάξει, πρέπει να περιορίσουμε όμω ε, τον χρόνο μιλίας ε, των βουλευτών ε, στο ένα λεπτό. Καθώ λυπάμαι πολύ, αλλά ήδη έχουμε καθυστερήσει και μετά έχουμε και ψηφοφορίε. Πρέπει κάπως να συντομεύσουμε. Παρακαλώ, κύριε Γκόμε. Σα ευχαριστώ πολύ για την δουλειά που κάνετε, για τις συστάσει σα και για τον προβληματισμό που θέτετε. Πραγματικά είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και δεν ακολουθούνται οι συστάσεις σα, Αλλά δεν είστε μόνο και εμεί κάνουμε συστάσει που δεν ε, ε, ακολουθούνται. Ο ειδικό ε, απεσταλμένος ε, του ΟΗΕ στη Λιβύη τον περασμένο μήνα μα είπε ότι οι Υπουργοί Εσωτερικών έχουν πολύ στενόμυαλη αντιμετώπιση ε, ότι υπάρχουν σημαντικέ απειλέ ε, προ την Ευρώπη και γι' αυτό και δεν ακολουθούνται αυτέ οι συστάσει. Και όχι μόνο είναι παράδεκτο που η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει ε, αυτά τα κέντρα κράτηση και τα αποκάλυψε και ο ίδιο κέντρα κράτηση στη Λιβύη, αλλά και κατάρτιση για την οποία πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακτοφυλακή. Κανεί δεν παρακολουθεί ποιε είναι οι προεκτάσει. Και ουσιαστικά εκείνοι τι κάνουν, πυροβολούν τους μετανάστες κάθε φορά που ε, πρέπει να εξηγήσουν τι συμβαίνει με τα ε, πλοία του Ιταλικού ναυτικού. Είναι γελίο που έρχονται κάποιοι και μας λένε για μια εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής με το ίδιο σκεπτικό, με αυτή την αισθενόμυαλη προσέγγιση των Υπουργών Εσωτερικών που δεν καταλαβαίνουν το διακύβευμα εδώ. Και πραγματικά είναι κάτι παραπάνω από γελίο. Είναι απαράδεκτο και εγκληματικό σαν στάση. Η κυρία Σπινέλη έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβουλευτικό Φόρουμ για αυτή την έκθεση και έχω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, και συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε η συνάδελφος προηγουμένως, σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, παρακολούθησης και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλείται να μην ε, εκπαιδεύσει, να μην καταρτήσει την Λιβική ακτοφυλακή δεδομένης ε, της άστατης ε, κατάστασης των Λιβικών θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να υποστηρίξει την κατάρτιση της λευκής ακτοφυλακής. Επομένως, υποθέτω ότι η Frontex δεν μπορεί να έρθει σε αντίθεση με το Συμβούλιο σε αυτό το σημείο. Υπάρχει λοιπόν εδώ μια σημαντική αντίφαση. Αυτό είναι το πρώτο. Μετά, κάτι το οποίο πραγματικά με ανησυχεί. Χθες ανακοίνωσαν οι Ιταλικές αρχές την πρόθεσή τους να παρεμποδίζουν τα σκάφη χωρίς Ιταλική ή Ευρωπαϊκή σημαία που προσπαθούν να μπουν ε, ε, να σταθμεύσουν, να δέσουν μάλλον στους Ιταλικούς λιμένες. Ουσιαστικά τα σκάφη των ΜΚΟ έτσι σκάφη τα οποία καθημερινά μας ε, στέλνουν και μαθαίνουμε μάλλον ε, ε, τα γεγονότα με τα πλοία που βυθίζονται και το καθεξής. Όμως πλέον δεν υπάρχει ουσιαστικά συντονισμένη ανταπόκριση έρευνας και διάσωσης. Θα ήθελα λοιπόν και τη δική σας γνώμη ως προς αυτήν την κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου, εδώ υπάρχει κίνδυνος σοβαρής ε, παραβίασης του θαλάσσιου δικαίου και της ανθρώπινης ε, σύμβασης ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Άντρουσον. Ευχαριστώ πολύ <laughs> για την έκθεση. Θα ήθελα Επίση και εγώ ε, να πω ότι είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση και αυτά τα, αυτό το, αριθμητικό στοιχείο που αναφέρατε σήμερα. 2.005 άνθρωποι πατέχασαν τη ζωή τους. Κάποιοι βλέπουν αυτόν τον αριθμό και νομίζουν ότι είναι χρονολογία ή ένα απλό στατιστικό στοιχείο. Ε, και όχι άντρες, ε, γυναίκες, μικρά παιδιά που πνίγηκαν στη θάλασσα σε αυτό το υγρό νεκροταφείο που είναι πλέον η Μεσόγειος. Και οχι άντρε, γυναικες μικρα παιδια που πνιγηκαν στη θαλασσα σε αυτο το υγρο νεκροταφειο που ειναι πλεον η μεσογειος και θελω πραγματικά και εγώ ανασημεριστώ την απόλυτη ε, αγανάκτηση που εξέφρασαν και άλλοι συνάδελφοι. Είναι πολύ ανησυχητικό ε, αυτό που αναφέρει η έκθεσή σας για τις ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις εθνικές συνοριοφύλακες και την αστυνομία. Και αυτό συνεχίζει να υπάρχει ως κατάσταση και στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Frontex, πιο συγκεκριμένα στη Βαλκανική. Τι μέτρα λοιπόν υιοθετούνται για, την, για να αποφευχθούν τέτοιου είδους ζητήματα καταστρατήγησης του ε, διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρει ε, η έκθεσή σας, ιδίως ό,τι αφορά τα ουγγρικά και σερβικά σύνορα. Ξέρω ότι έχει ήδη αναφερθεί, αλλά πρόσφατα ακούστηκαν ε, πολύ ανησυχητικές ε, αναφορές ε, ότι δηλαδή οι λιβικές αρχές πυροβολούν ε, ε, κατά σκαφών που διασώζουν πρόσφυγες. Έχουν ληφθεί μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτών των προσφύγων και των σκαφών διάσωσης. Χαιρετίζω επίσης ε, τις ε, επιφυλάξεις ε, που θέτεται για τη συνεργασία με την Τουρκία. Η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Παρότι ε, χθε βγήκαμε από ένα τρεμερή διάλογο και υπήρξαν κάποιες αναφορές εκεί για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Βλέπετε ότι ιδίω στην Ελλάδα λέγεται ότι θα πρέπει να νομοθετήσει και να τους αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα. Ενώ σαφώς και επανειλημμένος και ρητός ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πει ότι η Τουρκία δεν είναι ασφαλής χώρα. Μας λένε όμως ότι ιδίω εξαιτία τη τρέχουσα κατάσταση ε, στην Τουρκία ε, για τα, με τα θεμελιώδη δικαιώματα και εφόσον όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι ε, ασφαλής χώρα ούτε καν για τον ίδιο τον πληθυσμό, πόσο μάλλον για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, γι' αυτό θα ήθελα να επαναλάβω την άποψή μα ότι δεν θα πρέπει να επιστρέφονται μετανάστες και πρόσφυγε προ αυτή τη χώρα. Ξέρω ότι ε, πιέζει ο χρόνος. σα ευχαριστώ που μα δώσατε τη δυνατότητα να θέσουμε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ. Να σα ενημερώσω ότι θα πρέπει, εάν θα περνήσουμε περισσότερο χρόνο στο θέμα αυτό, να... Ε, αναβάλουμε το επόμενο, διότι δεν θα προλάβουμε να τα συζητήσουμε επαρκώς. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε σύντομοι. Ένα λεπτό. Ξέρω, είναι πολλά που θα πρέπει να υποθούν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι εξαιρετικά σύντομη. Αλλά ίσως πρέπει να δώσουμε τον ίδιο χρόνο ομιλία σε, σε όλους ε, τους αγορητές, προσθέσω να μείνω όμω ένα λεπτό. Αρχικά να σα ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή τη ετήσια έκθεση που είναι ιδιαίτερα εμπιστευτομένη και ήταν και πολύ καλή παρουσίασή σα. Γιατί και από τον κανονισμό του Frontex αναφέρεται ότι το συμβουλευτικό φόρουμ πρέπει να έχει πραγματική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Πρώτο, πολύ γρήγορο ερώτημα. Έχετε όντω ε, απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα, σε όλα τα στοιχεία, σε όλους ε, ε, σε όλες τι τοποθεσίε όπου υπάρχουν πρόσφυγες ή υπάρχουν προσκόμματα και τι είδους προσκόμματα είναι αυτά. Γιατί ακούμε διάφορα ε, για ψευδείς πληροφορίες, fake news που ε, μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές και μπορούν να επηρεάσουν αυτά τα στοιχεία που πρέπει να είναι πραγματικά ακριβή ε, και αντικειμενικά. Δεύτερον, μιλήσατε για απαράδεκτες ε, και απάνθρωπες συνθήκες ε, διαβίωσης ε, των μεταναστών και των προσφύγων, ιδίως στην Ελλάδα. Οι συνάδελφοί μας μετέβησαν πρόσφατα στην Ελλάδα. Έχουν υπάρξει προσπάθειες βελτίωσης αναφέρεται. Εσεί Εσείς συμμερίζεστε αυτή την άποψη ή σε ορισμένα μέρη και πιο συγκεκριμένα στα νησιά είδατε τέτοια ιδιαίτερα στοιχεία. Μετά. έχετε ένα πρόγραμμα που λέγεται Vega Children. Θεωρώ ιδιαίτερα ανησυχητική ε, την κατάσταση για τα χιλιάδες παιδιά και σε ε, σωματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Για όλα αυτά τα παιδιά λοιπόν ε, που κάποια βέβαια χάνουν και τη ζωή τους, αλλά άλλα έχουν αυτό το τραύμα ε, τελικά, πώς όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στο πρόγραμμα αυτό. Η κυρία Βεργιά, αλλά και πάλι μόνο για ένα λεπτό παρακαλώ, γιατί ήδη είστε η τρίτη ομιλήτρια της ομάδας σας. Συγγνώμη που ανήκουμε σε μια πολιτική ομάδα για την οποία είναι τόσο ανησυχητικό αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ τον κύριο Κέσλε. Γνωριζόμαστε από καιρό και πραγματικά εκτιμώ τον τρόπο με τον οποίο ε, μας παρουσιάζει τη δουλειά που κάνει. Εγώ δύο σημεία θέλω να επισημάνω. Ο μηχανισμός ε, ενστάσεων ε, και ένα θέμα στο οποίο έχουμε πολύ μεγάλο ρόλο να δραματίσουμε, γιατί η τήρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας δικηβεύεται εδώ. Ιδίως εκτίμησα και αυτό που είπατε ε, για την αμφισβήτηση των ΜΚΟ και για τις ανησυχητικές αναφορές ε, σε ό,τι αφορά τον Frontex και από ό,τι βλέπω νομίζω ότι έχει διευθυνθεί τα πράγματα και χαίρομαι. Ελπίζω να ξεπεράσουμε, να περάσουμε και στις πράξεις, όχι μόνο στα λόγια. Συμφωνώ με αυτά που αναφέρθηκαν για την Τουρκία και για την κατάρτιση ε, της Λιβικής Εκτοφυλακής. Ένα σημείο προβληματισμού, πέρα και τα όσο είπε η Ναταλή Γκρισβέκ, για, την, για τις προεκτάσεις της συμφωνίας με την Τουρκία, γιατί βλέπω ότι ο λένε και μεγαλύτερος αριθμός ε, ευάλωτων ατόμων ε, μένει, ξεμένει μάλλον στα ελληνικά νησιά. Έχετε πληροφορίες πώς νομίζετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση και θα ήθελα να μας ε, παρουσιάσετε περισσότερο την ανησυχητική κατάσταση ε, στα ουγγροσερβικά σύνορα γιατί οι δικές μου πληροφορίες μου αναφέρουν ο πρόεδρος διακόπτη. Ναι, ένα λεπτό κύριε πρόεδρε. Ε, για την Frontex. Μεταξύ τη Frontex και της Ουγγρικής αστυνομίας. Η Frontex ε, ουσιαστικά εκμεταλλεύεται και κρύβεται πίσω από τις ε, κακές πρακτικές που ακολουθεί και η Ουγγρική αστυνομία. Ευχαριστώ κυρία Τσινίτσι. <clears throat> Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Απλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλευτικού Φόρουμ του Frontex, όχι μόνο για την έκθεση, αλλά για την καθημερινή τους εργασία για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς του οργανισμού Frontex, διότι μιλάμε για την αξιοπρέπεια ανθρώπων και αυτό θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα πάνω απ' όλα. Η κυρία Σπινέλη αναφέρθηκε στην ανησυχητική κατάσταση στην Ιταλία. Η Ιταλία κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει ζωές. Και νομίζω ότι ε, προσέχει ιδιαίτερα τους ανηλίκους. Μιλήσατε για τη σωστή κατάρτιση εντός του Frontex ε, και αυτό χρειάζεται για την προστασία των παιδιών. Ε, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, να ζητήσω να μου δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει κάποιο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των παιδιών και γενικά των πιο ευάλωτων ομάδων που έχουν πέσει θύματα βίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νετφέλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κέσλερ για την παρουσίασή σας. Ομολογώ ότι παρότι ε, αισιόδοξη από τη φύση μου, ε, ε, νιώθω απελπισία. Οι κυβερνήσεις των κρατών μελών μιλάνε για θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό όμως είναι το χαρτί περί πολιτικών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι γραφειοκρατική διατύπωση ε, για κάτι που ουσιαστικά κρύβει την πραγματικότητα, που είναι πολύ διαφορετική. Έχω μια ερώτηση. Ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση. Αναφερθήκατε στην εκπαίδευση της ακτοφυλακής στη Λιβύη και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λένε «Α, πολύ ωραία, ναι, εμείς τους διδάσκουμε ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα». Ίσως ε, εγώ να φταίω, αλλά είμαι πολύ καχύποπτη στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Κάστερ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας αυτή, καθώς και για την ε, αφοσίωσή σας ε, στο θέμα αυτό. Ε, Φέτος 2.005 ε, άνθρωποι έχουν πνιγεί στην ε, Μεσόγειο, πέρσι πάνω από 5.000 άνθρωποι. Ε, εγώ βρίσκω ότι είναι τροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διάσωσης. Φαίνεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυριαρχεί η ιδέα ότι η Μεσόγειος είναι μια ζώνη απειλαγμένη από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πόσες μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, ασχολούνται με τη διάσωση ανθρώπων στη Μεσόγειο. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Σύμφωνα με αναφορές, οι μη κυβερνητικέ αυτές οργανώσεις ε, αναζητούν επαφή με σκάφη του Frontex ε, και τα σκάφη αυτά δεν αντιδρούν σε περίπτωση που οι μη κυβερνητικέ οργανώσει λένε ότι είναι ήδη υπερβολικά φορτωμένα τα σκάφη του και δεν μπορούν να σώσουν άλλους. Ε, εσείς γνωρίζετε τέτοια περιστατικά όπου τα σκάφη της Frontex να αγνοούν εκκλήσεις για βοήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους ευρωβουλευτές ε, και θα ήθελα να σας καλέσω να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Αποφασίστε εσείς μεταξύ σας ποιος θα απαντήσει. Σας παρακαλώ όμως να παραμείνετε εντό του χρόνου. Ευχαριστώ. Μακρύ ο κατάλογος των ερωτήσεων. Θέλω να επενθυμίσω ότι η εντολή του συμβουλευτικού μας φόρουμ είναι πολύ περιορισμένη. Συνεπώς δεν έχουμε εντολή να σχολιάσουμε τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, για παράδειγμα. Δεν έχουμε εντολή να σχολιάσουμε άλλα πολιτικά αντίστοιχα ζητήματα. Όμως σημειώνω τα δικά σας σχόλια, αλλά δεν ε, μου επιτρέπεται να σχολιάσω. Όσον αφορά την κατάρτιση της Λιβικής Ακτοφυλακής, δεν νομίζω ότι εμεί ξέρουμε περισσότερα από εσά. Προς το παρόν και εμείς έχουμε μια σαφή εικόνα για το ποιος σχεδιάζει να κάνει τι και με ποιον. Ακούσαμε ότι θα υπάρξει κατάρτιση και για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνει αυτό και ποια ακριβώς θέματα θα συμπεριληφθούν σε αυτήν την κατάρτιση, υπό ποια μορφή κλπ. Κατά τη δικιά μου προσωπική άποψη το πράγμα πηγαίνει ακόμα πιο μακριά. Ακόμα και αν υπήρχε μια εξαιρετικά καταρτισμένη λιβική ακτοφυλακή, τι θα γινόταν με τους πρόσφυγες αυτούς που έπιανε η ακτοφυλακή και μετά βρίσκονταν υποκράτηση εκεί. Το θέμα πάει πιο μακριά δηλαδή από το ζήτημα της Λιβικής ακτοφυλακής. Όσον αφορά κυρώσεις, Ιταλία, για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις κλπ. Ε, τώρα τα μαθαίνω κι εγώ αυτά. φαίνεται πάντως να αντιβαίνει στην επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Frontex στην επιστολή τους έχουν πει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία κατά καμίας μη κυβερνητική οργάνωσης που προβαίνει σε διασώσεις στη θάλασσα ότι έχουν ε, πέσει σε κάποιο αδίκημα. Συνεπώς, οποιασδήποτε κυρώσεις σε βάρος μιας τέτοιας μη κυβερνητική οργάνωσης δεν έχει βάση. Για το θέμα των Βαλκανίων και την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα στα Βαλκάνια είναι ένα πολύ καλό θέμα για το οποίο συνεργαζόμαστε με τη Frontex. Πρώτα απ' όλα για διευκρινήσεις το ποιος είναι υπεύθυνο γιατί σε αυτές τις χώρες και ποιος ελέγχει ποιον όπως επίσης για το ποια θα ήταν η κόκκινη γραμμή για τη Frontex προκειμένου να αποσυρθεί. Ακόμα δεν έχουμε οριστική απάντηση. Οπότε συνεργαζόμαστε με την Frontex επ' αυτού, αλλά προς το παρόν δεν είμαι σε θέση να σας δώσω αρκετές πληροφορίες για την Ελλάδα. Αναφερθήκατε στην έκθεσή μας μετά από επίσκεψη στην Ελλάδα το 2016. Και επιτρέψτε μου εδώ να το ξεκαθαρίσω. Δεν ήταν για να ελέγξουμε πώς έχει η κατάσταση συνολικά στην Ελλάδα. Ήταν απλώς μία επίσκεψη για να, έχουμε, να συλλέξουμε πληροφορίες για το πλαίσιο μέσα στο οποίο δράει η Frontex στην Ελλάδα. το φόρου μας δεν είναι το σώμα που μπορεί να ελέγξει τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και κυρίως στα νησιά. Σημερίζομαι όμως τις ανησυχίες όσον αφορά την κατάσταση στα νησιά, ότι δεν είναι καλή. Ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους και η συνάδελφος θα απαντήσει για το θέμα των ε, παιδιών και τα άλλα. Ευχαριστώ Στέφαν. Εγώ θα απαντήσω για την πρωτοβουλία όσον αφορά την προστασία των παιδιών της Frontex. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σαν στόχο να εντοπίζει τα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν στα αεροδρόμια τα ευρωπαϊκά. Και το Συμβουλευτικό Φόρουμ κλήθηκε από τη Frontex ως ε, παρατηρητές προκειμένου να συμμετέχουμε στη δράση αυτή για τρία χρόνια. Και το 2016 όντως εντοπίσαμε 13 ή μάλλον όχι. Συμμετείχαν το 2016 13 από εμά στη δράση αυτή και ασχοληθήκαμε με δύο πράγματα. Με τον ε, εντοπισμό και το δεύτερο ήταν η οικοδόμηση ικανοτήτων, δηλαδή στα αεροδρόμια πώς θα βοηθήσουμε να εντοπιστούν τα παιδιά αυτά που βρίσκονται σε κίνδυνο. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων με εμπειρογνώμονες, με την ακτοφυλακή, με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, οπότε είναι μια, ένα καλό παράδειγμα συνεργασίας της Frontex με το φόρου μας. Και με χαρά διαπιστώσαμε ότι η Frontex χρησιμοποιεί την ίδια ιδέα και όσον αφορά τα χερσαία σύνορα. Και μάλιστα έχει προχωρήσει πιο πολύ. Στηρίξαμε τη Frontex και σε αυτό. Και ολοκληρώνεται τώρα αυτή η πτυχή. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα βρείτε στη σελίδα, την ιστοσελίδα της ε, Frontex. Τώρα, αυτό που ρωτήσατε εσείς, κυρία, για την ε, κατάρτιση για την προστασία των παιδιών. Έχουμε στηρίξει την Frontex για να ετοιμάσει κατευθυντήριες γραμμές, τα είπε και ο Στέφαν, το οποίο λέει πώς μπορούν να υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, κατάρτιση των αξιωματούχων που δρούν στα σύνορα. Έχουμε και ενισχύσει το σκέλος που έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε συμπεριλάβει όλος ιδιαίτερο τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες. Αυτή είναι μία πτυχή λοιπόν σχετικά με την οποία στηρίξαμε τη Frontex. Επιπλέον, το είπε και ο Στέφαν, ότι έχουμε εκπονήσει μελέτη για την προστασία των παιδιών με συστάσεις. Αυτό είναι κάτι βέβαια που ενημερώνεται και συνεχίζεται. Η Frontex είναι εκείνη πάντως που έχει την εντολή να φροντίσει για κατάρτιση όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Οπότε το δικό μας φόρου, το συμβουλευτικό, θα την στηρίξει τη Frontex εφόσον ζητηθεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μας δώσετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε την έκθεσή σας μαζί σας. Έχει μοιραστεί σε όλους τους ευρωβουλευτές μας και προσβλέπουμε σε επόμενη συνάντηση. Τώρα, γιατί είμαι αυστηρός με το χρόνο ομιλίας και θα συνεχίσω. Είναι ότι μπορεί να μην έχουμε ψηφοφορίε, αλλά έχουμε τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη ακόμα που πρέπει να τα ξεπετάξουμε σε μία ώρα. Οπότε, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο του διερμηνείς, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε σύντομοι και να περιοριζόμαστε σε ένα ή δύο λεπτό καθένας. Να τηρείτε το χρόνο σας λοιπόν παρακαλώ για να μπορέσουν όλοι Τώρα, επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ανταλλαγή απόψεων, Παρουσίασε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ολοκληρώνης Διαχείρισης των Συνόρων και αυτό στα πλαίσια του κανονισμού για την διαχείριση των συνόρων. Είμαστε σε διαδικασία προκειμένου να εκπονήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση των συνόρων, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει. Η Digi Home είναι εδώ, ο κύριος Καλοτσέντσκι, ο οποίος θα ενημερώσει την Επιτροπή μας για την δομή που προβλέπεται και για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας αυτής και τι θα συμπεριληφθεί στη στρατηγική αυτή και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική. Έχετε 10 λεπτά το πολύ. Παρακαλώ και μετά θα πάρουν το λόγο οι ευρωβουλευτές για ερωτήσεις, σχόλια κτλ. Πείτε μας αν θέλετε το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Παρακαλώ. Uh, Καλημέρα και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε μια γενική επισκόπηση σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Συνόρων Δεδομένων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της διαδικασίας αυτής, είναι πολύ σημαντικό για μας ε, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα στην αρχή της διαδικασίας για να κάνουμε αυτή την παρουσίαση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Εφόσον η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου θα είναι ε, ζωτική σημασία για την όλη διαδικασία. Δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε θα διατρέξω εν συντομία το ιστορικό υπόβαθρο. Δεν μιλούμε για κάποια νέα έννοια. Η ευρωπαϊκή ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων είναι μια έννοια που υπάρχει εδώ και καιρό στην Ευρώπη. Το 2002 ήδη υπήρξε μια ανακοίνωση με ορισμένες συστάσεις. Μετά το 2006 το Συμβούλιο ε, προσδιορίσε αυτή την έννοια βάσει του μοντέλου ε, ελέγχου συνόρων, τα πολύ συγκεκριμένη και σημαντική εξέλιξη στην συνθήκη της Λισαβόνας, υπάρχει διάταξη που λέει ότι σταδιακά θα πρέπει να βελτιώνουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων στην Ευρώπη. Βέβαια, Πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αυτή πέρσι όταν ε, υιοθετήθηκε η Ευρωπαϊκή, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός ε, ε, για την ακτοφυλακή και συνοριοφυλακή που έθεσε τις βασικές έννοιες και προϋποθέσεις της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων και για πρώτη φορά ενεργοποίησε αυτή την έννοια στη συνθήκη. Υπενθυμίζω ότι βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής βασιζόμαστε σε ένα ε, πρότυπο ελέγχου τεσσάρων επιπέδων ε, που έχει να κάνει με μέτρα στις τρίτες χώρες, με τις γειτονικές τρίτες χώρες, μέτρα ε, συνοριακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα, αλλά και μέτρα εντός της ζώνης Σέγγεν. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι διευκρινίζεται στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή, ε, διευκρινίζονται οι θεσμικές ε, ευθύνες ε, για την πραγματική εφαρμογή αυτής της έννοιας. Επομένω, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή αναλαμβάνουν το καθήκον της πραγματικής και αποτελεσματικής υλοποίησης. Και εδώ έχουμε βέβαια και τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής, αλλά και της, ε, την ακτοφυλακή και τη συνοριοφυλακή ε, στα κράτη-μέλη. Αυτό πάντα θα πρέπει να γίνεται ε, σε ένα πλαίσιο μεκτή αρμοδιότητας και ευθύνης. Εξίσου Σημαντικό είναι το γεγονός ότι στον κανονισμό προσδιορίζεται ένας ε, κατάλογος 11 στρατηγικών στοιχείων. Στο άρθρο 4 μπορείτε να βρείτε και τους ορισμούς ε, που είναι πολύ ε, πιο ολοκληρωμένοι από πλευρά περιεχομένου. Θα ήθελα μόνο να επισημάνω ότι από πλευρά Επιτροπής Υπάρχουν και κάποια οριζόντια στοιχεία που σίγουρα θα πρέπει να λεφθούν υπόψη όταν μιλούμε για την επιχειρησιακή διάσταση και την ολοκλήρωση της διαχείριση των συνόρων και για την ανάπτυξη στρατηγικών. Ιδίω εδώ έχουμε κατά νου τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν σε όλα αυτά τα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για την κατάρτιση και την έρευνα και ανάπτυξη, που δεν αναφέρονται ρητός εδώ, αλλά ε, έχει συμφωνηθεί ότι απλώς ε, διέπουν το όλο σύστημα οριζοντίως. Τώρα, για τη στρατηγική διαδικασία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για να γίνει επιχειρησιακή αυτή η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων που προβλέπεται στον κανονισμό, στην τρίτη έκθεση προόδου για την ε, εφαρμογή της ακτοφυλακής και ε, συνοριοφυλακής του Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε ένα πολύ συγκεκριμένο και ε, φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα και μία στρατηγική, η οποία θα πρέπει να παρτίζεται από τρία παράλληλα στοιχεία κατάρτιση μια τέτοια στρατηγική σε πολιτικό επίπεδο τα θεσμικά όργανα, μετά υιοθέτηση μια τεχνικής και επιχειρησιακής στρατηγικής από τον Οργανισμό τη Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακή και Συνεργοφυλακή και τρίτο επίπεδο θέσπιση εθνικών ε, στρατηγικών ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων σε όλα τα κρατημέλη. Σκοπός ε, τη διαδικασία, προτινόμενο σκοπό, από πλευρά τη Επιτροπή είναι η επίτευξη ενός ενιαίου επιχειρησιακού πλαισίου για την οργανωμένη διαχείριση συνόρων που θα ισχύει συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή στην Ευρωφυλακή για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της έννοιας. Ορισμένα στοιχεία για αυτά τα επιμέρους στοιχεία της διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Στρατηγική λοιπόν, για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συνόρων, IBM, που θα συμφωνηθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Προκύπτει από μια ξεκάθαρη αναγκαιότητα πολιτικής καθοδήγησης για τη θέσπιση ε, αυτού του πλαισίου. Αναφέρεται στην λογική σκέψη 8 του κανονισμού ότι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι ευθύνη των ενωσιακών θεσμικών οργάνων. Ταυτόχρονα είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει και στενή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό και στην Επιτροπή είμαστε σε στενή συνεργασία με τον Frontex για αυτό το σκοπό. Πρόθεση της ε, στρατηγικής αυτής είναι η θέσπιση ενός ε, πλαισίου πολιτικής που θα εντοπίσει στόχους και προτεραιότητες και θα θεωρείται ουσιαστικά περισσότερο ε, πολιτική διακυβέρνηση ε, καθοδήγηση και όχι μιας πολύ συγκεκριμένη στρατηγική επιχειρησιακού χαρακτήρα. Γιατί αυτό προβλέπεται για το δεύτερο ε, επιμέρους στοιχείο που προανέφερε και θα αναφέρω και στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, η Επιτροπή θέλει να υιοθετήσει μια ανακοίνωση ε, που στοχεύουμε να δημοσιεύσουμε τον Οκτώβριο του 2017. Βέβαια, τα θεσμικά όργανα αυτά τα οποία θα διαμορφώσουν αυτή την ε, πολιτική στρατηγική είναι όμως πολύ σημαντικό να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Κομισιόν και Συμβουλίου. Και βέβαια η Κομισιόν στην προετοιμασία, κατά την προετοιμασία της ανακοίνωσης θα βρίσκεται σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τα θεσμικά όργανα. Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι εφόσον αυτή η διαδικασία θέλει την θέσπιση αυτού του πολιτικού πλαισίου από όλα τα ενωσιακά θεσμικά όργανα, η Κομισιόν θα καλέσει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετήσουν και να προσυπογράψουν αυτή την ανακοίνωση. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη διάσταση, το δεύτερο επιμέρου στοιχείο που ανέφερα, στο άρθρο 3.2 του κανονισμού για την ακτοφυλακή και στην αναφέρεται ρητός ένα βασικό νέο καθήκον για τον οργανισμό, θέσπιση τεχνικής και επιχειρησιακής στρατηγικής για την οργανωμένη διαχείριση συνόρων. Εμείς θεωρούμε ότι έτσι πραγματικά έχουμε την επιχειρησιακή διάσταση αυτής της πολιτικής και εφόσον ε, η, διαδικασία, η όλη διαδικασία έχει ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει το στόμετρο δυνατόν να ξεκινήσουμε τις εργασίες σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και βέβαια τα κράτη-μέλη. Σε τελική ανάλυση όμως, η τελική υιοθέτηση του πλαισίου μπορεί να γίνει μόνο όταν υιοθετηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα η στρατηγική, η πολιτική στρατηγική. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που προβλέπετε και ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν όλα πάνε καλά, ενδεχομένως ε, να υιοθετηθεί η στρατηγική τον επόμενο Φεβρουάριο. Η τελευταία τώρα διαφάνεια που ήθελα να επισημάνω την τρίτη διάσταση αυτής της στρατηγικής θέσπιση εθνικών στρατηγικών διαχείρισης συνόρων από τα κρατημέλη. Μια ξεκάθαρη ε, προϋπόθεση από τον σχετικό κανονισμό. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχει μόνο σύσταση προς τα κρατημέλη όπως υπήρχε παλιά στο εγχειρίδιο της ζώνης Ένγκεν να υπάρχει με τη διαστρατηγική. Υπάρχει πλέον υποχρέωση θέσπισης τέτοια ε, στρατηγική. Οι στρατηγικέ των 100 μελών θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τεχνική και επιχειρησιακή στρατηγική που θα θεσπίσει ο οργανισμό και να λαμβάνουν υπόψη τα βασικά στοιχεία, ιδίω στο άρθρο 4 του κανονισμού. Και πάλι θα πρέπει παραλλήλου να ακολουθούνται αυτές τις διαδικασίες, όμως η Επιτροπή αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη τουλάχιστον μάλλον το αργότερο έξι μήνες μετά την υιοθέτηση της επιχειρησιακής στρατηγικής να ευθυγραμμίσουν και την εθνική του στρατηγική. Γιατί υπάρχουν τέτοια στρατηγικές σε κάποια κράτη-μέλη, κάποια άλλη κράτη-μέλη τις αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή Οπότε θα πρέπει έξι μήνες το αργότερο μετά την υιοθέτηση της στρατηγικής να υιοθετηθεί και αυτό το πλαίσιο. Και η Επιτροπή θα ήθελε ε, να αξιολογήσει μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης ΕΝΓΕΝ αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία με τα βασικά στοιχεία και σε πολιτικό και σε τεχνικό, επιχειρησιακό, στρατηγικό επίπεδο. Να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή ο οργανισμός ε, ε, παρέχει αρρωγή στα κρατη μέσω ε, του αντίστοιχου προγράμματος κατάρτισης IBM. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο ε, για την πραγματική εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Θα μείνω εδώ, δεν ξέρω πώς θα έχω πάει από πλευράς χρόνου. Αυτά όμως από μένα και με τα χαράς ε, να απαντήσω στις ερωτήσεις. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καλοτσίνσκι για την παρουσίασή σας αυτή. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στους ευρωβουλευτές για να ακούσουμε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Καταρχάς ε, θα δώσω το λόγο στη Ρομπέρτα Μετσόλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εκπροσωπώ εδώ τον Άρτης Πάμπριξ που ζητεί συγγνώμη που δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα εδώ, που είναι η πρώτη φορά που συζητάμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων στην Επιτροπή μας. Ο κανονισμός, ε, όπως μόλις είδαμε, καθορίζει τις βασικές αρχές. Το άρθρο 4 του κανονισμού αναφέρει 11 στρατηγικά στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν ε, τμήμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης ε, των συνόρων. Έλεγχη των συνόρων, συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ανάλυση κινδύνου, επιθεωρήσεις και έλεγχη και στη θάλασσα κλπ αναφέρεται ότι η ολοκληρωμένη αυτή στρατηγική αποτελεί ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο οργανισμός ε, έχει καθήκον να εφαρμόσει ε, τη στρατηγική αυτή και να συνδράμει τα κράτη-μέλη στην ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής αποτελεί απαραίτητο στοιχείο και σε μεγάλο βαθμό ε, θα ε, κριθεί η επιτυχία του μέσου αυτού. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο και προκλητικό έργο και ένα έργο με πολλές προκλήσεις και Κατά τις διαπραγματεύσεις υπήρχε σαφής ε, κατανόηση ότι το πολιτικό πλαίσιο θα πρέπει να δημιουργηθεί σε στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και γι' αυτό δεν ενδείκνεται να, ζητήσουμε, να ζητηθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο απλά να εγκρίνουν τη στρατηγική χωρίς τη δυνατότητα να συζητηθεί και να ε, συνεισφέρουν κατά τη διάρκεια τη διαδικασία Και γι' αυτό ο συναδελφός μου Άρτης και εγώ επικροτούμε το γεγονό ότι έχουμε επιτέλου αυτή τη συζήτηση εδώ στην Επιτροπή μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Η Πίρκε Τσίπελ, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τα όσα ήδη είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα. Ε, θα μπορέσω να είμαι σύντομη όσον αφορά το περιεχόμενο του ε, θέματος ε, της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ε, επιμείναμε ε, η ε, αναζήτηση και διάσωση να αποτελεί σημαντικό έργο του Frontex και επίσης να μιλάμε για παραπομπή των προσώπων που ζητούν διεθνή προστασία. Για όλα τα τμήματα της εντολής αυτής θα ήθελα να τονίσω αυτό που ήδη υπόθηκε, ότι θα πρέπει να διευκρινιστούν ε, τα στοιχεία αυτά στην πολιτική στρατηγική που θα αποφασιστεί από όλους τους νομοθέτες. Γι' αυτό θα ήθελα να επιμείνω το πρώτο βήμα να είναι ακριβώς η σωστή πληροφόρηση, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε ανταλλαγή απόψεων ώστε να αναδιοργανώσουμε την πολιτική μας στρατηγική που όχι μόνο να λαμβάνει υπόψη αυτό που μας παρουσιάστηκε αλλά η πολιτική στρατηγική αυτή να αναπτυχθεί και όλοι οι οργανισμοί να μπορέσουν να οργανώσουν και τις επιχειρησιακές στρατηγικές μετά από αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε και για αυτή την παρουσίαση. Έχω ορισμένα ερωτήματα γιατί θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά τεχνική η παρουσίαση. Και νομίζω ότι λείπει λίγο το περιεχόμενο. Ακούγοντάς σας έχουμε την εντύπωση ότι ε, και η ΜΕΝ και η ΔΕ περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αν κατάλαβα καλά, λέτε ότι οι εθνικές στρατηγικές θα πρέπει να υιοθετηθούν τελικά, όμως μέχρι τότε αρκετά κράτη-μέλη προβαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ολοκλήρωσης της ε, διαχείρισης συνόρων. Δεν ξέρω τελικά τι πλαίσιο θα διαμορφωθεί λοιπόν για αυτή τη διαδικασία, πώς θα πρέπει να εργαστούμε και στο πνεύμα αυτών που είπε η κυρία Σίπελ μέχρι τον Οκτώβρη Εάν περιμένουμε δηλαδή την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή περιμένουμε εμείς να πλαισιώσουμε κάπως από πλευράς περιεχομένου αυτή την ε, πολιτική διαδικασία. Να θέσουμε εμείς ένα πολιτικό περιεχόμενο στις κατευθύνσεις που μπορεί να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη στρατηγική. Thank you very much. And the next... Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. αναζήτηση και διάσωση είναι ένα από τα στρατηγικά στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων. Ε, αν ισχύει αυτό, θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ε, βλέπει την ανακοίνωση της Ιταλίας ε, την χθεσινή που δεν θα επιτρέψει επιτρέψει ε, την ε, αποβίβαση σε σκάφη ε, μη Ιταλικής σημαίας που ασχολούνται με την αναζήτηση και διάσωση. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις και παρατηρήσεις από τους Ευρωβουλευτές, θα δώσω πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας είναι κάποιες ε, πράγματι πολύ σημαντικές πρώτες σκέψεις. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι είναι σαφές ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως ε, στην διαδικασία αυτή. Αυτό αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Μαΐου κατά την προετοιμασία της διαδικασίας αυτής. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της διαδικασίας και έχει πραγματοποιηθεί μια τεχνική συνάντηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Μόλις όμως καθοριστούν πιο συγκεκριμένα τα διάφορα στοιχεία της στρατηγικής αυτής, ε, θα είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, διότι τέθηκε ερώτηση σχετικά με το πώς θα λειτουργήσουν στη διαδικασία οι εθνικές στρατηγικές. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη ε, είναι υποχρεωμένα να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης Schengen και μέσω άλλων μηχανισμών μηχανισμών, έχει καταστήσει σαφέ ότι είναι απόλυτα απαραίτητο κάθε κράτος μέλος να έχει μια στρατηγική. Τώρα πια είναι κιόλα κιόλας κάτι τέτοιο. Ε, διάφορα κράτη-μέλη έχουν λάβει και σχετικές συστάσεις από τον Μηχανισμό Αξιολόγησης σε ΒΑΛ. Ο κανονισμός απαιτεί από τα κράτη-μέλη Ε, να ε, συμμορφώνονται με την ε, στρατηγική και με τις συστάσεις. Πολλά λοιπόν ήδη έχουν εκπονήσει στρατηγική. Πρέπει λοιπόν τα κρατη να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής. Και για μας είναι σαφές ότι μια πολιτική στρατηγική είναι απαραίτητη ότι είναι απαραίτητο να δώσουμε κατευθυντικές γραμμές σχετικά με το τι μορφή θα πρέπει να έχει ε, μια εθνική στρατηγική. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει. Παρουσιάσαμε το χρονοδιάγραμμα μετά από την υιοθέτηση της στρατηγικής ολοκληρωμένης ε, διαχείρισης. Ε, πρόκειται όμως για ένα θέμα που απαιτεί πολύ συντονισμό και συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι η αναζήτηση και διάσωση πράγματι αποτελεί ένα στρατηγικό στοιχείο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρόκειται για θέμα το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Δυστυχώς ε, δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω την κατάσταση στην Ιταλία. Φαντάζομαι ότι ο εκπρόσωπος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δώσει πληροφορίες ε, σε σχετική συνέντευξη τύπου. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε έτσι αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Θα πραγματοποιηθεί τεχνική συνάντηση των εμπειρογνωμόνων κάποια στιγμή μέχρι τον Σεπτέμβριο και κατόπιν θα εκδοθεί η ανακοίνωση της Επιτροπής το πιθανότερο τον Οκτώβριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή υπόψεων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης πάνω στην κοινή ανακοίνωση για νέα όθηση της εταιρικη σχεσης σχέσης Αφρικής-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ε, γνωμοδοτήσει πάνω στην έκθεση της ε, ΔΕΒΕ και η συντάκτρια της νομοδότησής μας ε, είναι η κυρία Κέγκε. Η Επιτροπή μας θέλει να ακούσει σχετικά με το σημείο 5.1 γ της ανακοίνωσης διαχείριση της ε, μετανάστευσης και κινητικότητας. Ε, θα ήθελα πρώτα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και κατόπιν θα δώσω το λόγο στους ευρωβουλευτές που θα τον στήσουν ε, συμπεριλαμβανομένης της εισηγητής. Δίνω λοιπόν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Where your colleagues sit with the Commission. so Ευχαριστώ. Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση έρχομαι, Διευθυντρία για την Αφρική. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις βάση τη ανακοίνωση που φαντάζομαι έχετε δει και βέβαια το θέμα είναι το μεταναστευτικό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα Πραγματικά μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα να σας δώσω μία εικόνα ε, της ε, Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Δεύτερον, ε, σε τι επικεντρωνόμαστε όταν εξετάζουμε τη διαχείριση των συνόρων και την κινητικότητα. Και μετά να κάνω και μια σύντομη επισκόπηση των εμβληματικών πρωτοβουλίων που έχουμε προτείνει στην ανακοίνωση. Αν δείτε πρώτα την Σύνοδο Κορυφής, όπου η μετανάστευση θα είναι ένα κέριο σημείο, σκοπός μας είναι να δώσουμε πραγματικά μια όθηση, αν θέλετε, ε, για μια πολιτική, ένα πολιτικό μήνυμα. Είναι σύνοδος κορυφής, επικεφαλής λοιπόν αρχηγή κρατών και κυβερνήσεων από την Αφρική και την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα συνεδριάσουν για να συνομιλήσουν για το μέλλον αυτής της συνεργασίας. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει ένα ε, θετικό μήνυμα γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη Ε, έχουν ηγετικό ρόλο στους περισσότερους ε, τομείς συνεργασίας. Το κεντρικό μέλημα είναι η επένδυση στην νεολαία. Και γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε και αυτή την θετική κατεύθυνση. Έχουμε δύο βασικές ε, οδούς που επισημαίνουμε και στην ανακοίνωση. Θέλουμε να οικοδομήσουμε πιο ανθεκτικά κράτη και κοινωνίες που συμπεριλαμβάνει ζητήματα συγκρούσεων, ε, συστημάτων διακυβέρνησης και μετανάστευσης, που θα, στα οποία θα σταθώ εγώ σήμερα. Υπάρχει και μια άλλη άγουσα που συνδέεται με τη ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίω για τους νέους. Αν δείτε το δεύτερο θέμα που ήθελα να θίξω, ε, διαχείριση της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Εμείς θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα... Η μετανάστευση, δηλαδή κινητικότητα, είναι εξαιρετικά ε, σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με την οικονομία, την ασφάλεια και την κοινωνία και στην Αφρική και στην Ευρώπη. Και φαντάζομαι ότι και εσείς ε, ως ευρωβουλευτές τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται λοιπόν να επισέλθω σε λεπτομέρειες για το πώς επηρεάζεται το πολιτικό προσκήνιο στην Ευρώπη. Σίγουρα όμως έχει να κάνει, σε μεγάλο βαθμό επηρεάζει και την πολιτική σκηνή στην Αφρική. Το πλαίσιο πολιτικής για μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, προσδιορίζεται ουσιαστικά στη διαδικασία της Βαλέτας, όπως ε, αναφέρεται, όπου έχουμε ουσιαστικά ένα σχέδιο δράσης. Τέσσερις είναι οι βασικοί πυλώνες αυτού του εγγράφου που μπορώ να σας παρουσιάσω στη συνέχεια αν θέλετε. Το σημαντικό ουσιαστικά είναι ότι συμπεριλαμβάνει την επένδυση στις ε, βασικές αιτίες μιλά για την ε, νόμιμη μετανάστευση, αναφέρεται στην ε, επιστροφή και επανεισδοχή, ε, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τα εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται στη μετανάστευση. Έχουμε λοιπόν μια ολιστική προσέγγιση που διαμορφώνει το τελικό πλαίσιο πολιτικής. Θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε τρία ζητήματα που θα δείτε και στην ανακοίνωση. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση σε περιφερειακό επίπεδο, Προφανώς ε, και πρόκειται για ανθρώπους δηλαδή που διέρχονται τα σύνορα και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Δεύτερον, θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το μερίδιο της ε, νόμιμης μετανάστευσης και κινητικότητας, να δούμε δηλαδή τη μετανάστευση και ως ε, μοχλό ανάπτυξης. Τρίτον, θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία για την παράτυπη μετανάστευση. Αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι θέλουμε μια σύνοδο κορυφής όπου θα τεθούν πολύ συγκεκριμένοι και απτοί στόχοι και παραδοτέα. Θέλουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε συγκεκριμένε εμβληματικές πρωτοβουλίες. Εδώ έχουμε δύο τέτοια στοιχεία. Πρώτον, να στηρίξουμε αφρικανικές πρωτοβουλίες για την ε, νόμιμη ε, ενδοαφρικανική μετανάστευση και ε, κινητικότητα και να αυξήσουμε την εργασια κατά των εγκληματικών δικτύων εμπορία ανθρώπων. Ειδικά το δεύτερο είναι αυτό που βλέπουμε από τότε που ξεκινήσαμε τις ε, εντατικές ε, διαπραγματεύσεις μετά τη Λεπεντούζα το 2015. Γιατί νομίζω ότι αυτό πραγματικά έφερε τα πάνω κάτω και από τότε αναπτύξαμε αυτό το σχέδιο πολιτικής που έχουμε αυτή τη στιγμή πλαίσιο πολιτική, Αμοιβαίο συμφέρον υπάρχει και για την καταπολέμηση ε, του, της ανθρώπων και της διακίνησης, γιατί πραγματικά αυτά τα χρήματα πρόκειται για πολύ σημαντικού πόρου, αλλά και για πολύ σημαντικά στοιχεία από πλευρά ανθρώπινων ζωών. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε ε, πολύ προσεκτικοί. Θα μείνω εδώ και αν θέλετε μπορώ να επισέλθω σε επίσης λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Is there any of your... Οι συναδελφοί σας μήπως από την Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ ή Home μήπως θέλουν και εκεί να πάρουν το λόγο. Όχι. Ωραία. Καλώς. Οπότε τότε το λόγο έχει η κυρία Κέγκε που είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησής μας. Και με το ποιος άλλος θέλει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχόλιά της. Ευχαριστώ και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τόσο μας είπε. Το 2017 θα είναι δίχως άλλο μια χρονιά αποφασιστική σημασίας για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Πρόκειται για δύο υπήρους που έχουν πολλά να κερδίσουν από αυτή τη σχέση και που πρέπει να ενισχύσουν και τις διμερείς τους σχέσεις, τις οικονομικές και τις πολιτικές. Αλλά έχουμε και πολλά να χάσουμε αν δεν δράσουμε. Από τη δικιά μας την πλευρά. Επιμένουμε πάρα πολύ στην ενίσχυση αυτή της εταιρική σχέσης. Οι σχέσεις της Ευρώπης με την Αφρική είναι βέβαια συχνά βασισμένες σε στερεότυπα, σε συσχετισμό δυνάμεων, οπότε καλά θα κάνουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την Αφρικανική Ήπειρο επίσης όρις, χωρίς να συμπεριφερόμαστε με πατερναλισμό. Ξέρουμε Κονγκό, Μαλή, εξακολουθούν να υπάρχουν συγκρούσεις, κοινωνική μιζέρια, αστάθεια, κάτι το οποίο δυστυχώς επηρεάζει την καθημερινή ζωή χιλιάδων ανθρώπων που ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή κάποτε. Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι σε τέσσερις χώρες, αυτό το έχουν πει και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο κίνδυνος είναι Λιμός, η Εμένη, Νότιο Σουδάν, Σομαλία για παράδειγμα, Μιλάμε για 20 εκατομμύρια ανθρώπους που κινδυνεύουν να πεθάνουν από λοιμό. Έπειτα, οι πληγές είναι τεράστιες. Η Αφρική όμως παραμένει μία ήπειρος γεμάτη δυνατότητες. Πρόσφατα μόνο αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τον πολιτισμό της Υπήρου αυτής. Ό,τι κενό λοιπόν πολιτικό παραμένει πρέπει να καλυφθεί. Δυστυχώς έχουμε αφήσει τους Κινέζους να δραστηριοποιούνται στην Αφρική, ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αραβική Χερσόνησο, που επενδύουν στην Αφρική σήμερα πολύ. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος δωρητής παγκοσμίω. Από τη δικιά μας την πλευρά πάντως να ξέρετε ότι θα επιμείνουμε στο θέμα της κινητικότητας, ιδιαίτερα με κάποια προγράμματα μέσω προγραμμάτων. Για μας είναι ζωτική σημασία και το θέμα της μετανάστευσης και για τις δύο επίρους. Έχουμε κοινή ευθύνη και έχουμε ευθύνη και από τη δικιά μας την πλευρά. Άρα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της αλληλεγγύης, να την εφαρμόσουμε. Και αυτό σε συνεργασία πάντα με την Αφρικανική Ήπειρο. Ξέρετε ότι εδώ βασιζόμαστε και στη διασπορά για επενδύσεις. Όλα πάντως πρέπει να γίνουν σε συνεργασία Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε επίσης ότι έχουμε πάρα πολλούς Αφρικανούς που έρχονται να ζητήσουν άσυλο στις χώρες μας, στην Ευρώπη. Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε σωστά, με κατάλληλες δομές υποδοχής στις χώρες όπου αυτοί φτάνουν. 12.000 έφτασαν στην Ιταλία πρόσφατα. Η Ιταλία λοιπόν χρειάζεται βοήθεια χρειάζεται αλληλεγγύη. Τις ευθύνε πρέπει να τις μοιραζόμαστε μεταξύ μας. Εξίσου. Πρέπει επίσης να δράσουμε και στην πηγή, δηλαδή να αποφύγουμε οι άνθρωποι αυτοί να κινδυνεύουν τη ζωή τους για να φτάσουν στην Ευρώπη. Και πρέπει να συνεργαστούμε με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες transit. Όλα αυτά αναφέρονται στο έγγραφο και ελπίζω να εγκριθούν και να δουν το φως της ημέρας κάποια στιγμή. Έχουμε ρεκόρ αφήξεις από την Αφρικανική Ήπειρο. Αν λοιπόν δεν καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ροές και αν συνεχιστούν οι ροές και στο εσωτερικό της Αφρικής αλλά και προς την Ευρώπη, αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Αφρική. Υπάρχουν και κάποιοι που μετακινούνται κατά ανάγκη. Οι αρχές του ΟΗΕ αποτελούν μια καλή βάση κίνησης. Πάντω, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εμεί από το δικιά μα την πλευρά πρέπει να επικεντρωθούμε στι αρχέ εκείνε που αναφέρονται στο ψήφισμα που μιλάει για μια συνολική προσέγγιση διαχείριση των ροών. Με την κυρία Μέτσολα η είναι συνεισηγήτρια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο για αυτό το θέμα. Η κυρία Λέχο και η κυρία Βερζάτ. Κανένα άλλο. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε Βαλέρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις αιτίες που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν την Αφρική και πηγαίνουν σε άλλες επίρους. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο δεν έχουμε τα εργαλεία για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να παραμείνουν, Διότι το θέμα εδώ δεν είναι η παράτυπη μετανάστευση, είναι η ακούσια μετανάστευση. Θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην ε, ακούσια και την ακούσια μετανάστευση. Έχουμε τους ανθρώπους που είναι φοιτητές, ερευνητές, ε, οι καλά εκπαιδευμένοι. Αυτοί θέλουν ε, να ταξιδέψουν, αλλά δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που καταφτάνουν. Σημαντικό είναι λοιπόν να ε, δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να καταλήψουν τη χώρα τους. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τη διάκριση αυτή. Αυτοί δηλαδή που εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή πρέπει και αυτούς που εγκαταλείπουν τη χώρα τους επειδή θέλουν. Διότι συχνά και οι δύο αυτές κατηγορίες ε, καταλήγουν να είναι παράτυποι μετανάστες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν νόμοι οδοί και για τους καλά εκπαιδευμένους, αλλά και για τους ανθρώπους που ε, δεν έχουν ε, ε, ανώτερα εκπαίδευση ή πιθανότατα δεν έχουν καθόλου εκπαίδευση. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε... εντός της δικής τους χώρας. Σημαντικό δηλαδή είναι να εξετάσουμε το σύνολο της αλυσίδας. Δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα άμεσα αν δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Αυτό θα απαιτήσει χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά και εμείς εδώ, να εξετάσουμε την νόμιμη μετανάστευση αλλά να φροντίσουμε να καλύπτουν όλα τα είδη των μεταναστών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο του κεφαλαίου για τη μετανάστευση. Επίσης, όταν μιλάμε για τη διασπορά, λέγει εδώ, ότι θα πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό της νόμιμης μετανάστευσης και κινητικότητας. Νομίζω ότι σαμποτάρουμε τον εαυτό μας. Διότι μιλάμε μόνο για αυτούς που ήδη βρίσκονται εδώ, αυτούς που ήδη έχουν καταφτάσει. Δεν μιλάμε για αυτούς όμως που στο μέλλον θα έρθουν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος ε, της ανάπτυξης ε, που θα βοηθήσει την Αφρική να ε, αναπτυχθεί με θετικό τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που μπόρεσα να συνεργαστώ με την κυρία Κίνγκε για την έκθεση αυτή. Γιατί πιστεύω ότι συμφωνούμε σε πολλά πράγματα. Τι έχω να πω. Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δώσει μια νέα όθηση στην εταιρική αυτή σχέση, αλλά έτσι και αλλιώς δουλεύουμε εκ παραλλήλου με την συνολική ε, προσέγγιση και με τον ΟΗΕ, οπότε και αυτή η εταιρική σχέση πρέπει να γράφεται σωστά με τα άλλα δύο στο ίδιο πλαίσιο. Πρέπει να έχουμε πράγματι μια συνολική προσέγγιση απέναντι στη μετανάστευση. Και το λέω για άλλη μια φορά. Όταν κοιτάμε τα νούμερα της μετανάστευσης, έχουμε 60 εκατομμύρια που είναι μετανάστες στον κόσμο και μόνο 35 εκατομμύρια Αφρικανοί. Και όταν βλέπουμε τα νούμερα επίσης, είναι η μετανάστευση από τον νότο στον νότο που αυξάνει και όχι αυτή από τον νότο στον βορρά. Αυτά είναι στοιχεία. Αν θέλουμε λοιπόν μια πραγματική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρικής και συμφωνώ με την κυρία Κίνγκη σε αυτό, πρέπει να υπάρχει πραγματικά εταιρική σχέση και να πάψουμε έτσι αποκαιοκρατικά να κοιτάμε την ε, Αφρική και να της λέμε τι πρέπει να κάνει. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα πρέπει να στηρίξουμε τη δημοκρατία, να σταματήσουμε να διαπραγματευόμαστε με δικτάτορες στο κέρας της Αφρικής, στο Σουδάν, στην Ερυθρέα. Θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια από αυτού. Εταιρική σχέση λοιπόν χρειάζεται οικονομική που να ευνοεί την ανάπτυξη και που να μην ευνοεί τις πολυεθνικές, τις ευρωπαϊκές ή άλλες ή τοπικών δικτατόρων να υπάρχει πραγματική κινητικότητα, ανταλλαγέ μεταξύ των δύο επίρων. Πρέπει να ανοίξουν όντω νόμιμε δίωδοι για την μετανάστευση και για του πρόσφυγε, αν θέλουμε να μην έχουμε πια πνιγμού στη Μεσόγειο. Να σταματήσουμε να έχουμε έμονη ιδέα με την παράνομη μετανάστευση. Εντάξει, θα υπάρχει και θα υπάρχουν και νεκροί στη Μεσόγειο όσο δεν υπάρχει νόμιμη μετανάστευση που να επιτρέπεται που να έρχεται από την Αφρική. Να σταματήσουμε επίσης να βάζουμε όρους στις συμφωνίες επανεισδοχής, να σεβόμαστε τα όσα έχουν υποσχεθεί οι χώρες επίσης για την αναπτυξιακή βοήθεια. Όσο η βοήθεια της διασποράς θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη των ευρωπαϊκών χωρών, τόσο θα συνεχίζουμε να περπατάμε ανάποδα. Ευχαριστούμε πολύ και ο κύριος είπε ότι έχει θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω. Μια καλή βάση για καλές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αφρική είναι το δίκαιο εμπόριο. Στο παρελθόν, στην εμπορική πολιτική ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αφρικανικές χώρες, εφαρμόζαμε πολιτική προς όφελος της ε, Ευρώπης και εις βάρος της Αφρικής. Να σας θυμίσω την ε, συμφωνία ε, όπου γεωργικές ότι γεωργικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταστρέψει οι αφρικανικές αγορές. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πορεία και να εφαρμόσουμε εμπορική πολιτική που να λαμβάνει υπόψη περισσότερο το συμφέρον των αφρικανικών χωρών και να διαμορφωθεί η πολιτική προς όφελος των αφρικανικών χωρών. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη μου παρατήρηση αφορά κάτι που ήδη υπόθηκε. Έχει να κάνει με τη μετανάστευση. Θα πρέπει να φροντίσουμε στο θέμα των ε, συμφωνιών ανάμεσα στη, σε χώρες της Αφρικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φροντίσουμε να αναφέρονται πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν αφρικανικά κράτη με δικτατορίες, ε, οι άνθρωποι προσπαθούν να διαφύγουν. Η τρίτη μου παρατήρηση είναι αυτό που είπε η συνάδελφος. Μεγάλο πρόβλημα στα αφρικανικά κράτη είναι συχνά πόλεμοι και εμφύλοι πόλεμοι. Ε, θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τις εξαγωγές όπλων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες της Αφρικής για να φροντίσουμε να υπάρχει η ειρηνική ανάπτυξη στην Αφρική. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μια σύντομη παρατήρηση της κυρίας Βαλέρο και μετά θα δώσω το λόγο στο, στην εισηγήτρια και στην Κομισιόν. Ναι, μια μικρή παρατήρηση, γιατί άκουσα ότι φαίνεται ότι είπα εγώ παράνομη μετανάστευση. Εγώ δεν χρησιμοποιώ ποτέ τέτοια λέξη. Μιλάω για μη εθελοντική, αναγκαστική μετανάστευση, παράτυπη ίσως, αλλά ποτέ δεν λέω παράνομη πρέπει να μιλάμε για σε εθελοντική βάση, μη εθελοντική βάση και να μην χρησιμοποιούμε ποτέ τον όρο παράνομη μετανάστευση, γιατί δεν υπάρχει παράνομη μετανάστευση και παράνομη μετανάστες. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ, ο Πρόεδρος. Κυρία Κέγκε, θέλετε να επανέλθετε. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα όσα είπατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το εκτιμώ ιδιαίτερα. Τώρα πρέπει να συνεργαστούμε για να ενισχύσουμε αυτή την εταιρική σχέση. Να υπενθυμίσω κάποια ραντεβού που μας περιμένουν. Είμαστε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έτσι δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε ότι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλάζουν κυρίως στα πλαίσια της Συμφωνίας Κοτονού και της περίοδου μετά τη Συμφωνία Κοτονού. Από τη δικιά μας την πλευρά πρέπει να δεσμευτούμε ώστε οι νέες αυτές σχέσεις να γραφούν σε ένα νέο νομικό πλαίσιο το οποίο θα μας οδηγήσει σε περιφερειακή προσέγγιση. Σήμερα πρέπει να κάνουμε προτάσεις για το τι θέλουμε να γίνει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μην ξεχνάμε δηλαδή, δεν υπάρχει μόνο το βραχυπρόθεσμο, αλλά και το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά τα πλούσια σχόλια που ακούσαμε και τις ερωτήσεις σας. Συμφωνώ απόλυτα όταν λέει η συγγήτρια ότι είναι η χρονιά της Αφρικής, ότι είναι αποφασιστικής ε, σημασίας. Ε, το 2017 πραγματικά για την Αφρική είναι ένας χρόνος ε, καμπή G7, G20 επικεντρώνονται στην Αφρική και θα υπάρξει και η δέσκευση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Πράγμα που σημαίνει ότι οι πλατφόρμες είναι πολυάριθμες για την Αφρική φέτος. Θέλω να θίξω τώρα διάφορα ζητήματα, αλλά να επικεντρωθώ κυρίως σε τέσσερα. <clears throat> Όσον αφορά την πραγματική, αυθεντική εταιρική σχέση, κάτι στο οποίο πολύ αναφερθήκατε. Αυτό ακριβώ είναι και στην καρδιά της ανακοίνωσή μας. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που για την Αφρικανική Ένωση το 2017 είναι και το έτος της νεολαίας, γιατί έτσι στρέφεται προς το μέλλον. Η εταιρική σχέση πάντως Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής συμπεριλαμβάνει σαν κύριο ζήτημα ακριβώς αυτό και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε στην πολιτική μας απέναντι στην Αφρική. Για την ε, ολιστική συνολική προσέγγιση. Πολλοί το ανέφεραν. Μα αυτό, όταν εγώ αναφέρθηκα στο πολιτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμεθα, το είπατε κι εσείς τι κάνουμε ασχολούμαστε με την νόμιμη μετανάστευση, με την προστασία των μεταναστών. Εδώ είναι που επισέρχεται και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα δίκτυα εγκληματιών. Συγγνώμη, πνίγηκα, λέει ο ομιλήτρια. <clears throat> Sorry. <clears throat> Migration is a touching... Ναι, η μετανάστευση, βλέπετε, είναι κάτι που όλους μας ε, αγγίζει, οπότε... Ωραία, θα προσπαθήσω να ξαναβρω τη φωνή μου και να επανέλθω. Ωραία. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά συνεχίζω. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι όταν μιλάμε για αυτή την συνολική ε, προσέγγιση για μετά το κοτονού, αν κοιτάξουμε την ίδια τη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής, ποια είναι η φιλοδοξία είναι να διασφαλίσουμε ότι οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων θα ασχοληθούν με τα ζητήματα της Αφρικής σε αυτή την ε, διάσκεψη και να προσθέσω και το εξή Πολύ αναφερθήκατε στη διασπορά και για τους σπόρους που έχουμε από την διασπορά σε σχέση με τους κρατικούς. Έχουμε διάφορα προγράμματα με τα οποία προσπαθούμε να εμπλέξουμε και τη διασπορά. Τώρα θέλω να ολοκληρώσω με το εξής κάτι που πάντα είχαμε υπόψη μας και όλοι αναφερθήκατε στους ανταγωνιστές μας, σε άλλους που δρούν στην Αφρική, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τη διαχείριση της μετανάστευσης. Αυτοί που μας έρχονται από την Αφρική και που μετακινούνται όλο και περισσότερο είναι κάποιοι τους οποίους πρέπει να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος. Όπως είπατε και πολλοί, πρέπει να υπάρχει πραγματικά μια πραγματική εταιρική σχέση και να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την μετανάστευση και με τους Αφρικανούς. Στην Αφρικανική πολιτική το θέμα της μετανάστευσης έχει μπει στην ατζέντα. Και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο. Τέλος, από τον Ιανουάριο, αν μη τι άλλο φέτος, το θέμα της διάσωσης και ε, της διόδου της κεντρικής Μεσογείου είναι κάτι για το οποίο συζητάμε πολύ. Δεν πρέπει, όταν μάλλον συζητάμε για τη μετανάστευση από την Αφρική, πρέπει να μιλήσουμε για την Λιβύη, για το 95% περνάνε από την Λιβύη. Γι' αυτό και πρέπει να δημιουργηθεί μια πολιτική λύση στη Λιβύη. Ναι, ξέρω είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά απλώς εδώ απαριθμίζω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και πώς αντιμετωπίζουμε συνολικά το θέμα της μετανάστευσης. Συνεπώς, κοιτάμε τις οικονομικές προπτικές, απασχόληση, δικαιώματα και διαχείριση της μετανάστευσης συνολικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι συγγνώμη που έχασα τη φωνή μου πριν, αλλά ξανάρχεται. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ, πολύ χαιρόμαστε για όλα αυτά. Καλό ήταν που σας είχαμε να ξέρετε ότι για την παρουσίαση της νομοδότησης της ΛΥΜΠΕ ε, από την κυρία Κέγκε προβλέπετε για την 31η Αυγούστου αμέσως μετά τις θερινές διακοπές που θα έχουμε έρθει ξεκούραστη. Θα αρχίσουμε συζητώντας αυτό το σχέδιο. Και με αυτά περνάω στο επόμενο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη που είναι και η αποστολή της Επιτροπής Λίμπε στη Europol 23 Μαΐου του 2017. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έστειλε την προσωπία για να επισκεφθεί τη Europol και συμμετείχαν στην αντιπροσωπή αυτή ο Άξελ Φως και ο κύριος Φως έχει ετοιμάσει μια έκθεση που θα μας παρουσιάσει τώρα. Έχετε το λόγο. Ähm, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η επίσκεψη στην Europol ήταν πολύ καλή και πολύ χρήσιμη και γι' αυτό ήταν κρίμα που μόνο εγώ ήμουν εκεί ως Ευρωβουλευτής. Ήταν δηλαδή μάλλον διμερής η επίσκεψη. Αυτό ήταν κρίμα. Θα ήθελα να καλέσω όσους ενδιαφέρονται για τέτοια θέματα να συμμετάσχουν σε τέτοιες επισκέψεις παρουσίαση που μας έκαναν εκεί ήταν πολύ εντυπωσιακή. Ενώ γνωρίζουμε τι κάνει η Europol, ήταν παρόλα αυτά λίγο διαφορετικό να το δούμε εκεί επί τόπου. Διότι ε, δύο-τρεις μέρες πριν ε, είχε εξαπλωθεί ο ιός I Wanna Cry. Και γι' αυτό ήταν ιδιαίτερα επίκαιρα τα θέματα αυτά. Είναι ενδιαφέρον επίσης να ακούσει κανείς τι ρόλο παίζει η Europol. Ασχολείται με το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ε, την διακίνηση ναρκωτικών, ε, το λαθρεμπόριο όπλων, ε, την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Έχουμε την συμφωνία Σέγγεν, Τρέβη. Ήταν πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά που είδαμε. Είχαμε δύο συνεδριάσεις ομάδας εργασίας. Το πρωί ασχοληθήκαμε με το ε, εμπόριο ανθρώπων, με την ε, διακίνηση ε, μεταναστών, ενώ το απόγευμα ασχοληθήκαμε με το κυβερνό έγκλημα. Ήταν λοιπόν χρήσιμα όλα αυτά. Δύσκολο είναι το θέμα της νομικής βάσης πάντα στη Europol. διότι είναι δύσκολο με διαφορετικές απαιτήσει τελικά να έχουμε κοινή δουλειά. Θα πρέπει αυτό να το προσέξουμε στο μέλλον. Η ίδια η Europol ασχολείται με το ότι το έγκλημα γίνεται όλο και πιο διασυνοριακό, όλο και πιο διεθνές. Συνεργάζεται λοιπόν και με τρίτες χώρες. Όταν θα έχει δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ΕΠΟ, και εφόσον και η Eurojust ε, πρικοδοτηθεί περισσότερο από την πλευρά μας, ε, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια συνδυασμού όλων αυτών. Ε, η Europol χρειάζεται επίσης περισσότερους εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο. Διαπιστώσαμε επίσης την τάση. Τα νομοθετικά και ρυθμιστικά μέτρα Τα μέτρα αυτά περιέχουν απαγόρευση για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Και έτσι έχουμε μεν εμπόδια στη δουλειά, χωρίς όμως αυτό να ε, επιφέρει βελτίωση της προστασίας των δεδομένων. Απλά καθυστερούν τα πράγματα. Επίσης, οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται τα κενά στις ε, ρυθμίσεις και γι' αυτό θα πρέπει προληπτικά να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Όσον αφορά τις μυστικές πληροφορίες. Και εδώ υπάρχει ένα κενό στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ήταν χρήσιμο και αυτό να επιληθεί. Επίσης, το θέμα των κοινωνικών μέσων δικτύωσης ε, και εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ερευνητικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Γενικά, υπάρχει επιθυμία για πιο ευέλικτες μορφές ερευνών. και ίσως ε, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα θέματα αυτά με το βλέμμα στο μέλλον. Όσον αφορά το έγκλημα, διαπιστώνουμε συνεχώς ότι εξαπλώνεται το έγκλημα ως υπηρεσία, crime as a service. Μπορεί κανείς δηλαδή να ε, ε, αγοράσει, να αναθέσει ή ε, να μισθώσει ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Είδαμε ότι έχουμε όλο και περισσότερες ε, κυβερνοεπιθέσεις όπως αυτή η τελευταία του I Wanna Cry με πολύ ευρία εξάπλωση και με τα bitcoins θα πρέπει να ασχοληθούμε. Δηλαδή γενικά με τον τομέα της πληροφορικής. όσον αφορά τη βιομηχανική κατασκοπία. Η Κίνα και η Ρωσία δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα στον τομέα αυτών. Ως νομοθέτες, αυτό συμπέρανα εγώ τουλάχιστον, θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τα θέματα αυτά. Αυτά ήταν τα συμπεράσματά μου θα ήθελα να σας συστήσω να ε, εξετάσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερη ομάδα να επισκεφτεί την Χάγη και αυτό δεν θα στοιχήσει υπερβολικά πολύ. Αξίζει τον κόπο να δείτε τα πράγματα αυτά επί τόπου. Ε, διότι προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε το έγκλημα σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις από πλευράς των παρόντων ευρωβουλευτών, από ό,τι βλέπω. Όχι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αξελφός, για την έκθεση αυτή και για την επίσκεψή σου στη Europol. Φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ημερησίας διάταξης. Θα ακούσουμε πώς έχει η κατάσταση όσον αφορά τον τριμερή διάλογο για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο. Ήταν ένα από τα πρώτα από τα σχετικά θέματα που ε, αποτέλεσε αντικείμενο τριμερούς διαλόγου. Πετύχαμε κάποια πρόοδο στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας. Ε, ο τελευταίος τριμερής διάλογος πραγματοποιήθηκε χθε το βράδυ και θα ακούσουμε από τον κύριο Νίτερ Μιούλερ τι πρόοδος έχει σημειωθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος χθε το βράδυ. Ο τριμερή διάλογο ε, επέτυχε μια ευρεία πολιτική συμφωνία σχετικά με τον, Ευρωπαϊκό Οργανισμό, τον κανονισμό και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Μετά από σχεδόν έξι μήνε διαπραγματεύσεων, η προκατακτική συμφωνία επετεύθηκε για τα 12 κεφάλαια τη πρόταση μεταξύ άλλων και για το πολύ ε, λεπτό ε, κεφάλαιο και νευραλική σημασία σε κεφάλαιο για τα προσωπικά δικαιώματα, δεδομένα και την τεχνική αρρωχή. Υπήρξαν σημαντικέ υποχωρήσει και από τι δύο πλευρέ, όμω ε, τελικά είναι καλές ισορροπημένη πρόταση. Θέλουμε πλέον να γίνει πλήρη οργανισμό ενωσιακό ο ΕΑΖΟ, αλλά να υπάρχει και ανεξαρτησία για, την, για να αυξήσουν τις ε, τεχνικές και επιχειρησιακές δραστηριότητε τους για να γίνουν θεματοφύλακας του Ευρωπαϊκού Κοινού Συστήματος Ασύλου ε, με πλήρη σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πετύχαμε αυτούς τους στόχους και τώρα θέλουμε να ακούσουμε από την πλευρά του Συμβουλίου ε, ποια είναι η γνώμη του για, αυτό, για αυτή την προσωρινή συμφωνία. Ταυτόχρονα, επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την ε, πολυθετική προσέγγιση, τη γραμματεία, τους κοιόδης ηγητές για τη στήριξή τους προς την προώθηση των διαπραγματεύσεων, ιδίως στο βράδυ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο για αυτό το σημείο. Θέλει κάποιο άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. σα ευχαριστώ και πάλι. Θα επανέλθουμε στις 2 το μεσημέρι με την κοινή ακρόαση ε, της Επιτροπής Λίμπα και της Επιτροπής Πέτη. Ευχαριστώ.